Καλησπέρα σας. Τα βασικά σημεία αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφαλείας Τροφίμων με την παρουσία του καθηγητού Σεραλίνη. Μετά θα ασχοληθούμε με την περιβαλλοντική επίπτωση των εγκαταστάσεων αιωλικής ενέργειας, την ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τη γνωμοδότηση για την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης υπάρχει και ένα λεπτό ζήτημα που έθεσαν συνάδελφοι, με βάση την απόφαση των συντονιστών να συζητηθούν τα σημεία 8 και 9 και κλεισμένων των θυρών. Θα ήθελα να εγκρίνετε την ημερήσια διάταξη ή, εν πάση περιπτώσει, να εκφράσετε αντιρρήσεις. Χάνκης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ αντιμετωπίζω προβλήματα με την ε, συνεδρίαση και κλεισμένο το θηρόν και θα ήθελα να σας θέσω και ένα ερώτημα σε σχέση με την, το τμήμα της συνεδρίασης που προτείνεται να είναι και κλεισμένο το θηρόν. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να είναι και κλεισμένο το θηρόν η εξέταση αυτά τα σημεία. Νομίζω ότι όλοι όσοι είμαστε παρόντες συμφωνούμε στο ότι ότι πρόκειται για ένα θέμα ιστορικού χαρακτήρα. Πρόκειται για μια διαφορά μεταξύ χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την επίλυση αυτού του προβλήματος θα πρέπει να εξασφαλιστεί μια συμφιλίωση μεταξύ των δύο χωρών, μια κατανόηση των αμοιβαίων επιχειρημάτων. Ο μόνος τρόπος για να γίνει κάτι τέτοιο είναι με την επικοινωνία, με το διάλογο και αυτός ο διάλογος θα πρέπει να είναι δημόσιος. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να αποτελεί μια ευρωπαϊκή αρχή ότι όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ανοιχτά και όχι κλεισμένο των θυρών. Αν λοιπόν υπάρξει ένα πρόβλημα το οποίο έχει ιδιαίτερα ευαίσθητο χαρακτήρα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και κλεισμένο από το θυρών. Μόνο στην κομμουνιστική εποχή γινόταν αυτά τα πράγματα στην Ουγγαρία. Αλλά τώρα έχει παρέλθει αυτή η εποχή. Και γι' αυτό εκφράζω την έκπληξή μου όταν βλέπω ότι ορισμένα θέματα προτείνεται να αντιμετωπιστούν ως ευαίσθητα και κλεισμένων των θυρών. Εδώ πρόκειται για ένα άτομο πάνω από 100 ετών που είναι αναφερόμενη. Είπε βέβαια ότι θέλει να έρθει εδώ. Δεν θέλει να νιώσει αυτό το οποίο θεωρεί ως ταπείνωση με την παρουσία της ε, εδώ. Ούτε και αυτό νομίζω ότι είναι φυσιολογικό. Μία οποιοδήποτε πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να θεωρήσει ταπείνωση μια τέτοια παρουσία. Συνάδελφε, Συνάδελφοι, για να εξοικονομήσουμε χρόνο θα ήθελα να πω ότι στην ημερήσια διάταξη και ιδιαίτερα σε σχετικές αποφάσεις τις οποίες προαναφέρθηκε η κυρία Χάνκης η Ολομέλεια αποφασίζει. Δηλαδή οι συντονιστές με βάση συγκεκριμένες πολιτικές ευαισθησίες πρότειναν μία συζήτηση και κλεισμένων των θυρών και αποφάσισαν με πλειοψηφία. Αλλά η Ολομέλεια της Επιτροπής αποφασίζει, χωρίς λοιπόν να παρατείνουμε τη συζήτηση, θα πρέπει να προτείνουμε κάτι άλλο για να προχωρήσουμε με τις εργασίες μας. Δεν θα ήθελα παρά να λάβουν το λόγο οι συνάδελφοι που το ζήτησαν. Θα ήθελα να είσαστε ιδιαίτερα σύντομοι, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Έχω να σας υποβάλω μια πρόταση. Προτείνω αυτό το οποίο προτάθηκε για την συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών να αποσυρθεί από τον αρμόδιο συντονιστή. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ανοιχτή η συνεδρίαση για τα θέματα αυτά. Φυσικά εναπόκειται στην Επιτροπή να αποφασίσει βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 49. Εδώ πρόκειται για στοιχεία εμπιστευτικά που έχουν να κάνουν με υπεράσπιση ενώπιον δικαστήριου. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να γίνει χρήση των συνεδριάσεων και κλεισμένων των θυρών. Αλλά εφόσον βρισκόμαστε σε μια κοινοβουλευτική συνεδρία, όπω είπε και η κυρία Χάνκη, εφόσον το δέχονται και οι άλλε πολιτικέ ομάδε, σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό να έχουμε ανοιχτή συνεδρία. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω να ψηφίσουμε υπέρ του να γίνει ανοιχτή συνεδρία. Νομίζω ότι θα πρέπει να ε, διασαφηνίσουμε κάτι, να διασαφίσουμε κάτι. Η Επιτροπή αναφορών δεν είναι ένας οργανισμός ειρήνης επί της γης. Δηλαδή δεν μιλάμε για εθνικές σειράξεις οι οποίες διαρκούν μία εκατονταετία. Εδώ έχουμε να κάνουμε με θέματα αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Αναφορών και μιλάμε για τα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν ισχύει αυτό που προαναφέρθηκε. Θα, καταλαβαίνετε, θα καταλάβετε λοιπόν γιατί οι συντονιστές ήταν απόλυτα σωστοί και συνετοί όταν είπαν ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί και κλεισμένων των θυρών, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Αναφορών δεν θα πρέπει να αποτελέσουν αρένα συζητήσεων ε, εσωτερικής κατανάλωσης καθαρά. Γι' αυτό αυτό το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί και κλεισμένο των θυρών. Και σας υπενθυμίζω ότι αυτή η απόφαση ελήφθη με την υποστήριξη όλων των συντονιστών ε, εξ ονόματος της πολιτικής τους ομάδας δηλαδή. Σας ευχαριστώ. Μαρβάτη. Ευχαριστώ. Αυτή η αρχή της και η αρχή της διαφάνειας είναι βασικές αρχές. Πρόκειται περί ανθρωπινών δικαιωμάτων εν Και για το ότι θα πρέπει εδώ να κατησχίσουν οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου. Δεν θα πρέπει να γίνει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επομένω, εν προκειμένου, πρόκειται να τα συζητήσουμε. Αυτά τα ζητήματα που είναι τόσο σημαντικά και δεν υπάρχει κανεί λόγο αυτό να γίνει και κλεισμένο. Το αντίθετο, για λόγου ε, δημοκρατική ούτω υπήρνη θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση του κοινού. Ακριβώ. Και η εμπειρία μου, η προτέρα, λέει ότι σε περιπτώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχή των προσώπων που, που, που, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται. Α πούμε, υπάρχει εδώ πέρα αυτή η κυρία 100 ετών, πόσο είναι, 101. Ε, είναι γνωστή η ιστορία τη, οπότε θα πρέπει να είναι εφικτό να μπορέσει να παραστεί. Πρόκειται για πραγματικά υπαρκτά πρόσωπα για την ζωή τους. Έτσι θα καταλάβουμε τι έχει γίνει και, και, και αν συντρέχει περίπτωση παραβίαση των δικαιωμάτων. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται ε, με ανοιχτή συνεδρίαση. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, λέει ο Πρόεδρο. Κύριο Γιάρ, μετά εσεί δεν θα λάβει άλλο το λόγο γιατί δεν είναι δυνατόν να αρχίσουμε συζήτηση επ' αυτού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας υπενθυμίσω την συμβιβαστική λύση που πετύχαμε στη συνεδρία των συντονιστών και να σας ζητήσω να την υποστηρίξετε. Κάναμε μια εκτανέστατη συζήτηση ε, για τα θέματα αυτά. Είπαμε ότι θέλουμε να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Είπανε πολλοί ότι δεν είμαστε αρμόδιοι για το θέμα αυτό. Είπαν άλλοι, αλλά μα είναι ένα πρόβλημα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να το συζητήσουμε. Υπήρξε δυσκολία λοιπόν να καταλήξουμε σε αυτήν την συμφωνία, τη συμβαστική, να συζητήσουμε μεν το θέμα αυτό, αλλά και κλεισμένων των θυρών. Θα ήθελα να πω στους συναδέλφους που ζητούν ανοιχτή συνεδρίαση να τους ζητήσω να μην ρίξουν το μωρό μαζί με τα ύδατα του μπάνιου από το παράθυρο, γιατί έχουμε μια συμβαστική λύση την οποία δεχτήκαμε όλοι και περιλαμβάνει τη συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών και εγώ θεωρώ ότι είναι μια καλή λύση. Δεν θέλω να ανατραπεί από την Επιτροπή μας. Εάν λοιπόν ε, θέλετε να υπάρξει μια ομαλή συζήτηση πρέπει να υποστηρίξουμε την συμβαστική αυτή λύση που ζητά να γίνει και κλεισμένο το θηρόν συζήτηση αυτού του συγκεκριμένου θέματος. Έχετε το λόγο, ναι. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, να έχω το λόγο να σας πω ότι διαφωνώ με αυτά που είπε ο Ρουμάνος συνάδελφος. Εγώ νομίζω ήταν εύστοχη η απόφαση Κάτι άλλο εδώ. Δεν πρόκειται για επίλυση διαφοράς μεταξύ Ουγγαρίας και Σλοβακίας. Πρόκειται περί διαφοράς μεταξύ του Σλοβακικού κράτους και Σλοβάκων πολιτών. Είναι σοβαρό θέμα και οι Σλοβάκοι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν πώς θα φτάσει σε μια απόφαση η Επιτροπή μας. Βεβαίως και σέβομαι τη γνώμη του κυρίου Γιάρ. Σέβομαι τα όσα έκριναν οι συντονιστές μας. Όμως, σας επισημαίνω ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πάρα πολλού κόσμου. Δεν είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει μόνο τους Ούγγρους και του Σλοβάκους έχει ευρύτερη σημασία για όλη την Ευρώπη. Άρα αυτό θα πρέπει εδώ πέρα να το ζητήσουμε συστηματικά, σε ανοιχτή συνεδρίαση. Όχι εν κρυπτό και απαραβίστο. Τίποτα δεν θέλουμε να κουκουλώσουμε. Uh, Ευχαριστώ. Μπορώ να είμαι πάρα πολύ σύντομη γιατί νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει αποφασιστεί είναι ήδη επαρκές και ζητώ από όλη την Επιτροπή να δεχτεί την απόφαση των συντονιστών σχετικά. Um, Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα είμαι σύντομος. ότι πρέπει να δείξουμε στους Ευρωπαίους ότι είμαστε 100% διάφανοι στις διαδικασίες μας και τέλο πάντων να κρυθεί η αποφασή μα μέσω ψηφοφορία στην Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή έχει γίνει. Το θέμα έχει εξαντληθεί. Το συζήτησαν οι συντονιστές. Κατέληξαν σε συμβαστική λύση οι συντονιστές για το πώς θα συζητηθεί. Είναι κρίμα. Η συνεδρίασή μας τώρα να γίνει ένα, ε, ε, ένα, ένα, μια πρόκληση της προεκλογικής για το Ουγγρικά κόμμα. Ακούσαμε επιχειρηματολογία από όλους και νομίζω ότι η θέση της Επιτροπής δεν είναι ομόφωνη. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις, και αυτό θα ήθελα να ρωτήσω από τους συναδέλφους μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν επί του θέματος αυτού. Θα ήθελα λοιπόν να συμμετάσχετε στην ψηφοφορία ιδιαίτερα ως προς την επιβεβαίωση της απόφασης των συντονιστών να διενεργηθεί η συζήτηση των σημείων 8 και 9 και κλεισμένων των θυρών. Διότι σας είπα ότι με βάση τον κανονισμό η Επιτροπή αποφασίζει. Δηλαδή, εγώ οφείλω να υποβάλω το θέμα στα μέλη της Επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν να ψηφίσετε υπέρ της απόφασης, σας παρακαλώ, καταρχήν ποιοι είναι υπέρ και όσοι βεβαίως είναι κατά θα καταψηφίσουν. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ της επιβεβαίωσης της απόφασης των συντονιστών να συζητηθεί αυτό το θέμα και κλεισμένων των θυρών. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 in favor. 9 υπέρ. Κατά παρακαλώ. Ποιοι είναι κατά. Μόνο 3, 4. 4 αντιτίθενται. Άρα η απόφαση της Επιτροπής ισχύει. Θα γίνει συζήτηση και κλεισμένων των θυρών. Θεωρώ λοιπόν ότι εγκρίνεται παράλληλα και η ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα στη συνέχεια να κάνω ορισμένες άλλες παρατηρήσεις. Στο σημείο 5 έχουμε την, μια πρώτη συζήτηση για τους ε, γενετικούς ε, τροποποιημένους οργανισμούς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σεραλίνη για την παρουσία του και να τονίσω ότι ο βασικός ετών, ο κύριος Μπράιαν Τζον, δεν είναι παρόν και μας απέστειλε δύο ε, γραπτές παρατηρήσεις. Θα παρακολουθήσει διαδικτυακά τη συνεδρίασή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, τον κύριο Μπέργμαν. Για τα σημεία 8 και 9 η Επιτροπή αποφάσισε να επιβεβαιώσει την ε, συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών. Αύριο θα είναι μαζί μας ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, ο κύριος Διαμαντούρος, ο οποίος ανακοίνωσε την παρέτησή του, υπέβαλε μάλλον την παρέτησή του, γι' αυτό και θα μας παρουσιάσει την τελευταία ετήσια έκθεσή του. Αύριο το πρωί η Επιτροπή θα λάβει υπόψη και την ετήσια έκθεση του κυρίου Μακμίλαν Σκοτ και θα ασχοληθούμε και με τη γνωμοδότηση του εισηγητή Τσίτσεστερ σε σχέση με την διπλή έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Επιτροπή ΑΦΚΟ έχει αναλάβει τη σχετική έκθεση. Μετά θα εξετάσουμε τις τροπολογίες της ε, έκθεσης του κυρίου Χούντι για, με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τέλος θα ασχοληθούμε με τις αναφορές της Γαλλικίας, την πρώτη της ε, Γαλλικίας και δεύτερης Μαδρίτης ως προς τις διερευνητικές επισκέψεις. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχουν, έχει εγκριθεί η ημερήσια διάταξη. το πρώτο θέμα. Ένα ερώτημα για την έκθεση σε σχέση με τη Γαλλικία. Κατά πόσο το έγγραφο για την αποστολή στη Γαλλικία θα δοθεί σε όλους τους συναδέλφους ή μονάχα στα επίσημα μέλη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής μας που πήγαν στη Γαλλικία. Γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι μόνο εγώ και η Τατιάνα έχουν το έγγραφο αυτό. Επειδή ήμασταν τα μέλη της αντιπροσωπείας, οι υπόλοιποι δεν ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Φαίνεται λοιπόν το θέμα αυτό θα έρθει σε συζήτηση αύριο, χωρίς να έχουν γνώση του εγγράφου οι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Τα έγγραφα θα έπρεπε να είχαν διανεμηθεί πράγματι σε όλα τα μέλη της Επιτροπής έτσι ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη συζήτηση. Εγώ μαθαίνω αυτή τη στιγμή ότι με βάση το αίτημα της κυρίας ε, μετά από έτοιμα της κυρίας Μπόλαντ, ε, τα έγγραφα δεν έχουν διανεμηθεί. Θα προσπαθήσω να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη και γιατί δεν έχουν διανεμηθεί αυτά τα έγγραφα τα οποία είναι απόλυτα, απολύτως απαραίτητα για την διενέργεια της αυριανής συζήτησης. Για να διευκρινίσω λιγάκι την κατάσταση αυτή. Όπως έλεγε ο κύριος Μπέρτμαν, η κυρία Βέρτμαν, συγγνώμη, χωρίς μικρόφωνο ο μιλητής. Ναι, ναι, συγγνώμη. Έλεγα ότι για να διευκρινίσω καλύτερα αυτό το οποίο έλεγε η κυρία Βέρτμαν εμείς δεν έχουμε τη μετάφραση στα ισπανικά. Νομίζω ότι μόνο αγγλικά υπάρχει αυτή η έκθεση που δεν είναι καν η γλώσσα του εισηγητή για το θέμα αυτό. Είναι κάποιες δυσκολίες που θα τις ε, εξηγήσει αύριο ο εισηγητής. Όλες αυτές οι τεχνικές δυσκολίες μας καθυστερούν. Εμείς θα θέλαμε να έχουμε ήδη το κείμενο της έκθεσης για να κάνουμε μια συζήτηση, αλλά η συγκή που σήμερα δεν έχουμε ακόμα την έκθεση στις διάφορες ε, γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ήμασταν στη Γαλλικία πριν από τρεις ή τέσσερις μήνες και ακόμα δεν έχουμε το έγγραφο μεταφρασμένο στις διάφορες επίσημες γλώσσες. Με όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη και σαν Προεδρείο και στη Γραμματεία. Όκεν. Μια μικρή παρατηρησούλα. Ε, είναι κάπως αφαίρετο να λέμε κάτι τέτοιο όταν ε, έχουμε μετάφραση σε όλες τις γλώσσες ή μετάφραση λιγότερες. και βλέπουμε να γίνει αναβολή στην πρώτη φάση και, με, και σε άλλες περιπτώσεις λέμε ότι δεν πειράζει. Είναι μια πρόφαση. Είναι μια πρόφαση που την επικαλούμαστε συχνά, αλλά μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα στα αγγλικά. Πόδος. Τα λαμβάνουμε και αυτό υπόψη και τώρα κλείνουμε με αυτό το σημείο. Το δεύτερο θέμα είναι η έγκριση των πρακτικών. Στις προηγούμενες συνεδρίες, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρώ ότι εγκρίνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. Όπως και σε κάθε συνεδρίαση σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει το παράρτημα σε σχέση με τις προτάσεις για τις αναφορές που έχουμε λάβει. Γι' αυτό μέχρι αύριο θα πρέπει να υποβληθούν. Διαφορετικά θεωρούμε ότι εγκρίνονται από την Επιτροπή όπως έχουν διανεμηθεί. Περνάμε λοιπόν τώρα στο θέμα υπαριθμών 5 της ημερήσιας διάταξης. το οποίο μας έχει απασχολήσει αρκετές φορές. Πρόκειται για τον αναφέροντα κύριο Μπράιαν Τζον, Βρετανικής Ιθαγένειας, σχετικά με τις ε, εικαζόμενες παραβιάσεις των γενικών αρχών που διέπουν τη δραστηριότητα της ε, Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των Τροφίμων σε σχέση με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Επίσης υπάρχει και μια δεύτερη της ε, Καρόλα Τουαντέλα και του, μια άλλη ε, αναφορά του κυρίου Μπράιαν Τζον γύρω από αυτό το θέμα. Όπως σας είπα, ο αναφέρον δεν είναι παρόν, γι' αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο στον καθηγητή, τον κύριο Σεραλίνη, για να μας πει ποια είναι η άποψή του επί του θέματος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι εδώ παρόν μεταξύ σας για να σας εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είμαστε αρμόδιοι ως ΕΦΣΑ τη στιγμή που υπάρχουν διάφορες συγκρούσεις συμφερόντων για το θέμα αυτό, ιδίω για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς αλλά και για τα παραστοκτόνα τα οποία συνδυάζονται με αυτούς τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Δημοσιεύσαμε ένα άρθρο τον προηγούμενο Σεπτέμβρη, το οποίο απορρίφθηκε από την ΕΦΣΑ και το βλέπετε εδώ στις διαφάνειες. Αυτό είναι ενδεικτικό του, τρόπου με τον οποίο οργάζεται η ΕΦΣΑ. Έχουμε 3 εκατομμύρια υπογραφόντων την ε, αναφορά μας και έχουμε επίσης 200 επιστήμονες σε μια άλλη αναφορά που ζητήσαν περισσότερη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ΕΦΣΑ και για τον τρόπο με τον οποίο απορρίπτει ορισμένα άρθρα και άλλοι 300 ε, επιστήμονες ζήτησαν να υπάρχει κατά αντιπαράθεση εξέταση των θεμάτων αυτών, κάτι το οποίο δεν έχει λάβει η χώρα. Είναι η μοναδική λοιπόν μελέτη αυτή που αφορά την ε, μακροχρόνια αξιολόγηση του Roundup, του, του πιο γνωστού παραστοκτόνου σε παγκόσμιο επίπεδο τις επιπτώσεις για τους εργαζόμενους στην γεωργία. Το Roundup είναι το πιο συνηθισμένο φυτοκτόνο σε παγκόσμιο επίπεδο. 80% των, των ε, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών είναι σχεδιασμένοι για να αντέχουν το Roundup, αυτό το παραστοκτόνο. Η ΕΦΣΑ είναι και διάδικος και δικαστής σε αυτή την περίπτωση γιατί έχει εγκρίνει τη χρήση αυτού του προϊόντος για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και έχει δώσει θετική γνωμοδότηση για το παραστοκτόν αυτό σε ό,τι αφορά την εμπορία αυτού του προϊόντος. Το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι ότι αν ζητήστε να μάθετε κατά πόσο το έγγραφό μας αυτό προς την ΕΦΣΑ ευσταθεί ή όχι, είναι σαν να του ρωτάτε αν η ΕΦΣΑ έκανε λάθος. Η ίδια η ΕΦΣΑ φυσικά δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι σφάλει. γιατί δεν έχουν λάβει υπόψη τους πολλούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία που δεν έλαβαν υπόψη τους ενώ θα έπρεπε να είχαν λάβει υπόψη τους. Σας υπενθυμίζω ότι η ΕΦΣΑ δεν ζήτησε πάνω από 90, από δοκιμές πάνω από 90 ημερών για, την, ε, για μία από τις ουσίες αυτές και επίσης για άλλες ουσίες οι οποίες βρίσκονται στα επιφανειακά ύδατα ή σε στοιχεία διατροφής. Το Roundup δεν περιλαμβάνει μονάχα το γλυφόσατο, αλλά και άλλες ουσίες. Εμείς έχουμε καταδείξει από το 2005 και εντεύθεν και είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο που δημοσιεύει για τα τοξικά χαρακτηριστικά του Roundup και τις επιπτώσεις του για τα ανθρώπινα κύτταρα και τα κύτταρα των θηλαστικών, έχουμε δημοσιεύσει πάνω από 12 άρθρα στον χώρο αυτό. Έχουμε εξετάσει τους μηχανισμούς που αποκαλούν τοξικότητα στα παραστοκτών αυτά και επηρεάσουν τα ανθρώπινα και τα ζωικά κύτταρα και έχουμε αντιμετωπίσει τα... Έχουμε εξετάσει τα αποτελέσματα που προκύπτουν για τους ανθρώπινους οργανισμούς. Ένας από τους κύριους κινδύνους λοιπόν των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών είναι τα υπολείμματα του ράουντα που παραμένουν μέσα στα τρόφιμα ή στα επιφανειακά ύδατα. Το έγγραφο αυτό απορρίφθηκε από την ΕΦΣΑ. Γιατί είπανε ότι δεν υπήρχαν αρκετά, αρκετές στατιστικές το γεγονός ότι το Roundup ε, σκότωνε περισσότερα θηλυκά ποντίκια από ό,τι την ομάδα ελέγχου. Όλα αυτά δεν τα δέχτηκε η ΕΦΣΑ. Το γεγονός επίσης ότι το Roundup δημιουργούσε πολύ περισσότερους καρκίνους στα θηλυκά ποντίκια από ό,τι σε, στην ομάδα ελέγχου. Θεωρήθηκε μη αποδεκτό αυτό από την ε, ΕΦΣΑ. Τα, η ομάδα ελέγχου έτρωγε τρόφιμα που δεν περιείχαν καθόλου γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και δεν είχαν καθόλου ε, Roundup. Είναι φανερό από τη μελέτη μας ότι το Roundup είναι υπέτειο για τα προβλήματα αυτά. Το πρόβλημα λοιπόν είναι η έλλειψη διαφάνειας. Έχουμε δώσει τα στοιχεία μας στα κύρια επιστημονικά περιοδικά με έλεγχο ομοτήμων σε παγκόσμιο επίπεδο, Food and Chemical Toxicology και περιμένουμε για πάρα πολύ καιρό να δημοσιευθούν. Η ΕΦΣΑ λοιπόν και η Μονσάντο, όλοι αυτοί οι οποίοι δεν δέχονται αυτό το έγγραφο, θα πρέπει να μας δώσουν πρόσβαση στα δεδομένα που χρησιμοποίησαν για την έγκριση αυτών των προϊόντων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους Ευρωπαίους πολίτες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τα οποία δικαιολόγησαν την έγκριση αυτών των προϊόντων για να ξέρουμε ποιος είναι πραγματικά έγκυρος και ποιος σφάλει σε αυτή την περίπτωση. Εμείς θέλουμε να έχουμε και τα αιματολογικά στοιχεία της μελέτης που έγινε για, τα, για να εγκριθεί η χρήση του Roundup. Είδαμε λοιπόν ότι, ότι το κλάφοσατ, η ενεργή ουσία, δεν είναι αυτή που προκαλεί την ε, τοξικότητα στα, ε, στους ε, ανθρώπους και στα ζώα. Η ενεργή ουσία που έχει τοξικό χαρακτήρα δεν είναι το γλαϊφωσάτ, αλλά είναι ένα άλλο στοιχείο της φόρμουλας του Roundup και το έχουμε δημοσίασει αυτό σε ένα άρθρο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι δεν υπήρξαν μέχρι στιγμής μακροχρόνιες αξιολογήσεις για την επίπτωση του Roundup. Έχουμε μονάχα τα στοιχεία της Άνσες, τα εμπιστευτικά στοιχεία του γαλλικού φορέα της Άνσες, που ήταν ακριβώς τα ίδια στοιχεία, τα οποία είναι όπως και αυτά της ΕΦΣΑ. Και η ΕΦΣΑ θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να αξιολογηθεί το Roundup σε μακροχρόνιο επίπεδο. Η Επιστημονική Επιτροπή της ΕΦΣΑ θεώρησε ότι δεν χρειάζεται μακροχρόνια αξιολόγηση των επιπτώσεων των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Για το NK603 δέχτηκε η ΕΦΣΑ να θέσει τα ακατέργαστα στοιχεία στο διαδίκτυο σε μορφή PDF που δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για στατιστική ε, μελέτη και η πνευματική ιδιοκτησία για τα θέματα αυτά, για το, τη μελέτη αυτή, ανήκε στη Μονσάντο. Αυτό το οποίο απέτρεπε τους ερευνητές από το να αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτή. Εμείς αξιολογήσαμε και πάλι τα στοιχεία αυτά και δείξαμε ότι υπάρχουν και αποτελέσματα για το σηκώτη και τα νεφρά των πειραματοζώων ε, μετά από μόνο 90 μέρες και πολύ πιο έντονα μετά από δύο χρόνια. Η ΕΦΣΑ αναγνωρίζει ότι είναι ανεπαρκή τα στοιχεία της Μονσάντο, αλλά τα έχουν δεχτεί. Βλέπουν ότι υπάρχουν σημαντικά αποτελέσματα, αλλά θεωρούν, όπως και η Μονσάντο, ότι δεν έχουν βιολογική σημασία. Εδώ υπάρχει ένας σημαντικός λόγος θεωρούν ότι τα ιστορικά στοιχεία των ποντικιών που ήταν ομάδα ελέγχου από το 1930 σε όλα τα εργαστήρια έχετε στοιχεία για τις ομάδες ελέγχου ώστε να μπορεί να έχει κανείς ιστορικά στοιχεία. Αλλά όταν δεν δημοσιεύονται ποτέ τα στοιχεία για τα αιματολογικά στοιχεία των ποντικιών δεν δημοσιεύονται αυτά ποτέ και όπως σας είπα η ΕΦΣΑ δεν έχει ζητήσει ποτέ μακροχρόνιες μελέτες και έχει δεχθεί ότι, ότι η σύνθεση των παραστοκτώνων μπορεί να μείνει απόλυτα εμπιστευτική. Βλέπετε εδώ λοιπόν τα αποτελέσματα του γλυφοσάτ το οποίο δεν είναι τοξικό γίνεται τοξικό μετά από την διάλυση σε διάφορες αγροτικές ουσίες που ραντίζονται το Roundup όμως είναι 10 φορές ή ίσως 100 φορές πιο τοξικό από το γλυφοσάτ. Αυτό όμως δεν γίνεται φανερό γιατί η ενεργή ουσία που οδηγεί στην τοξικότητα βρίσκεται μέσα στη φόρμουλα είναι πολύ εθιλοξικές ε, ενώσεις, το οποίο 15 που είναι σε πολλά φυτοκτόνα δεν υπήρξε ποτέ μελέτη για το θέμα αυτό, μελετήθηκε μονάχα στις, ε, στα κράτη-μέλη σε βραχυχρόνιο επίπεδο, αλλά δεν το έχει αντιμετωπίσει ποτέ σε μελέτη η ΕΦΣΑ. Και τα αιματολογικά δείγματα για το, τη μελέτη για το γλυφοσάτ είναι κλεισμένα σε ένα εργαστήριο και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα η ΕΦΣΑ να έρθει σε επαφή με αυτά τα ακατέργαστα, τα βασικά στοιχεία. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι το Roundup δημιουργεί προβλήματα στα, ευρυο, στα εμβριακά κύτταρα τα οποία ε, φωνεύει. Έχει δεχτεί λοιπόν η Επιστημονική Επιτροπή ε, την ε, μεταλλαγμένη πατάτα όταν μονάχα είχαν τραφεί με αυτήν πέντε ποντίκια κατά τη διάρκεια 90 ημερών. Ποιο λοιπόν είναι σε αυτό το παιχνίδι και ποιο είναι ε, ουσιαστικά. Έχουν τονιστεί οι συγκρούσεις συμφερόντων πολλές φορές στο Συμβούλιο της ΕΦΣΑ. Τα λεγόμενα ιστορικά στοιχεία που χρησιμοποιεί η ΕΦΣΑ όλα αυτά είναι ε, στρεβλά. Τα στοιχεία αυτά λοιπόν που μας λένε για τα ποντίκια αυτά και για τον έλεγχο του πόσους ε, όγκους μπορούν να δημιουργήσουν. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία είναι για ποντίκια τα οποία τροφοδοτούνται με δίαιτες οι οποίες δεν είναι γνωστό αν περιλαμβάνουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ή όχι. Επομένως τα στοιχεία αυτά τα ιστορικού χαρακτήρα μπορεί να έχουν και αυτά υπολείμματα από τόνα και γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Όλα αυτά τα κρύβει η, η ΕΦΣΑ με, τα με τη λεγόμενη εμπιστευτικότητα. Και ακόμα και οι ορισμένε άλλε ουσίε είχαν αποτελέσματα μέσα σε 90 ημέρε και η ΕΦΣΑ είπε ότι αυτό δεν ξεπερνάει το επίπεδο των ιστορικών στοιχείων. Η επιστημονική λοιπόν επιτροπή τη ΕΦΣΑ λέει ότι δεν ε, αυτό αποτελεί πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν 19 γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς που επανεξετάσαμε. Σε όλες τις περιπτώσεις τα όργανα τα οποία αντιμετωπίζουν τις τοξίνες, τα νεφρά και τα ε, σηκώτια είχαν προβλήματα. 42% των ε, παρενεργειών ήταν στα νεφρά. Ούτε και εκεί η ΕΦΣΑ δέχτηκε να κάνει μια ανεξάρτητη μελέτη για τα θέματα αυτά. Κλείνω λοιπόν, λέω ότι η ενεργή ουσία τοξικότητας του Roundup και ίσως για πολλά άλλα παρασιτοκτόνα σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους και τα φυλαστικά δεν είναι γνωστή. Το μόνο τέτοιο, η μόνη τέτοια ε, ουσία που γνωρίζουμε για τα φυτά δεν είναι κατά ανάγκη η πηγή τοξικότητας για τους ανθρώπους και τα θηλαστικά. Και η δεύτερη μου παρατήρηση είναι ότι δεν είναι διαθέσιμα τα ακατέργαστα στοιχεία, επιτρέπουν να χρησιμοποιούν τα λεγόμενα ιστορικά στοιχεία τα οποία δεν επιτρέπουν πραγματική ε, αντιπαράθεση γιατί ακόμα και αυτά τα ιστορικά στοιχεία προέρχονται από διατροφή με, με τρόφιμα τα οποία μπορεί να είναι μολυσμένα με μη με γενετικά τροποποιημένους ε, οργανισμούς. Γι' αυτό ζητήσαμε να υπάρξει άμεση παρουσίαση στο ίντερνετ για τα θηλαστικά που οδήγησαν στην έγκριση του Roundup. Αυτό δεν κοστίζει τίποτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-μέλη. Απλώς θα επιτρέψει στους διεθνείς εμπειρογνώμονες Όλοι οι επιστήμονες λοιπόν μπορούν να εξετάσουν τα στοιχεία αυτά από τη σελίδα του ίντερνετ και να δουν ποιο είναι το πρωτόκολλο το οποίο οδήγησε στην έγκριση των, ε, του Roundup από την ΕΦΣΑ. Αυτό θα δώσει δυνατότητα να υπάρχει δημοκρατία και διαφάνεια στην Ευρώπη για προϊόντα τα οποία μας αφορούν όλους αφορούν εμάς, τα παιδιά μας, όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Thank Ευχαριστώ καθηγητά Σεραλίνη. Ο κύριος Πέρμπεργκμαν έχει το λόγο. Παρακαλώ. Αγαπητοί βουλευτές, αγαπητή κυρία Πρόεδρε, η αυτό θεωρεί ότι είναι μια πάρα πολύ θετική ευκαιρία, ούτω ώστε να δούμε τι γίνεται με τη δημοσίευση του, της Σαραλίνη και των συνεργατών του. Αυτή η δημοσίευση έγινε πέρσι και επομένως έχει ως αντικείμενο να δούμε τι γίνεται με αυτή την τροφή που επί δύο χρόνια χορηγήθηκε σε αρουραίους για να δούμε τι γίνεται με αυτά τα, τα, τα, που περιέχουν αυτό την εν λόγω ενεργή ουσία. Και το συμπέρασμα της μελέτης ήταν ότι αυτοί οι τροπημένοι οργανισμοί και αυτές οι χημικές ουσίες ε, έχουν συγκέντρωση φυσικών ουσιών πολύ κάτω από τα προβλεπόμενα όρια και ήταν πάρα πολύ σοβαρά σε επιπτώσεις για τους αρρωίους αυτούς. Η ΕΦΣΑ έλαβε εντολή από την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ στις 26 Ενάτων, μία εβδομάδα αργότερα. Και ζητήθηκαν τα εξής πέντε τα οποία θα πρέπει επιγόντως να διεκπαιρεθούν. Η μελέτη να εξεταστεί πάρα πολύ προσεκτικά, να ζητηθούν διευκρινήσεις από τους συντάκτες, εάν χρειαστεί, να ε, ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν υπάρχουν νέα στοιχεία που έχει την μελέτη και ενδεχομένω να θεωρήσει ε, την απόφαση 603 η ΕΦΣΑ, εάν χρειάζεται να ληφθούν υπόψη οι προτάσει των κρατών μελών. Οι μελέτε ε, επικίνδυνοτητο σε συνεργασία με τι γερμανικέ αρχέ αλλά η Γερμανία ασχολείται με, το, με αυτό το glyphosate, το, κάτι το οποίο δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Advisory Forum ε, during the same week. Έγιναν αυτές οι επαφές, η ΕΦΣΑ ξεκίνησε την συνεργασία με το Συμβουλευτικό Σώμα, ούτως ώστε να ε, αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα και αυτό το Advisory Forum ε, έχει, απαρτίζεται από μέλη από τους ομολόγους μας όλη την Ευρώπη, από Ισλανδία και, και Ελβετία ακόμη, οπότε έτσι είμαστε εις θέση να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη με όλες το δυνατότητες, όλοι μαζί, να δούμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Είναι πιο σημαντική τουλάχιστον. Η ΔΕΦΣΑ δε εκάλεσε τα κράτη-μέλη να συζητήσουν το εγγραφό αυτό. Και Πολλοί είπαν ότι ήδη βρίσκονται οι εργασίες αυτές εν εξελίξη. Και συμφωνήθηκε ότι όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να αναλύσουν την ε, μελέτη από κοινού και να συγκρίνουν τα συμπράσματά τους ε, στην πορεία. Και αρχίσαμε λοιπόν μια σειρά από τηλεσυνεδριάσεις για να ανταλλάξουν πληροφορίες και έτσι να μπορέσουμε να συζητήσουμε την ερμηνεία των όσων ορίζει αυτή η μελέτη, να διεκπαιρεώσουμε ότι προβλήματα υπήρχαν. Και είχαμε έξι κρατημέλη τα οποία έλαβαν μέρο σε όλη αυτή τη διαδρομή και τη διαδικασία. Είχαν κληθεί όμω όλα τα κρατημέλη. Ζήτησε κατεπηγόντω να παράσχουμε συμβουλέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε εμεί είχαμε μια πολυκλαδική, διεπιστημονική ομάδα, τη συγκροτήσαμε και έτσι αναλύσαμε τη μελέτη αυτή σε δύο φάσεις. Πρώτα-πρώτα είχαμε ε, κάποιους από το πολιτικό μας και κάποιους ε, ειδικού σε δύο σε ε, πειραματικό σχεδιασμό, ε, τοξικολογία κλπ. Όλοι αυτοί κάνανε την αρχική ε, ανάλυση της μελέτης, αυτό έγινε και 4 δεκάτου έγινε σχετική δημοσίευση. Τόσο γρήγορα λοιπόν δεν είχαμε ενεργήσει για πάρα πολύ καιρό και αυτό το κάναμε, διότι θέλαμε να καλύψουμε τους στόχους της μελέτης, να καταλάβουμε τα στατιστικά μοντέλα και να μπορέσουμε να επισημάνουμε τυχόν κενά και μετά αυτά τα κενά να αρθούν. Δηλαδή να μπορέσουμε να, ζητήσουμε διευκρινήσεις από τους συντάκτες της ε, μελέτης και να μπορέσουμε να παράσχουμε πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μπορέσετε τώρα να καταλάβετε το το, το αυτής της δουλειάς ε, ε, καλέσαμε τους συντάκτες για να μπορέσουμε να συνοηθούμε γιατί θεωρήσαμε ότι έτσι θα καταλάβουμε πλήρως αυτό το οποίο χρειάζεται. Οπότε ε, το ανακοιμενό μας του κύριο Σαραλίνη του ζητήσαμε μέσα τον Οκτώβριο διευκρινήσεις και ήταν πάρα πολύ πολιτικό το ότι αυτή ότι, ότι ε, δεν, δεν, δεν συνεργάστηκε μαζί μας αρκετά. Παρά το ότι τα δική μας ήταν τα θέματα τα οποία απασχολούν τη δική μας υπηρεσία. Οπότε, 28 Νοεμβρίου δόθηκε τελική μας ανακοίνωση και καλύψαμε όλα όσα έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινιστούν και είπαμε ότι θα γίνει και κάποιο είδου ανεξάρτητη μελέτη και αξιολόγηση όλων αυτών τα κράτη-μέλη και αυτό έγινε χωριστά από Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Ιταλία και κάτω χώρες. Επίσης υπάρχει μια συνεχής αξιολόγηση για το glyphosate από τη Γερμανία. Και επίσης, λεφτική υπόψη, η απόκριση, η απάντηση τέλο πάντων ε, του Σαλήν και των συνεργατών του στις 9 Νοεμβρίου. Αυτό βέβαια αφορούσε τα περισσότερα από όσα είχαμε ρωτήσει, αλλά υπήρχαν και άλλα που είχαμε ρωτήσει, τα οποία μείναν αναπάντητα. Γι' αυτό σας λέω ότι θα έπρεπε να γίνει πιο σοβαρή προσπάθεια. Και αυτή η δημοσίευση δεν κάλυψε την, ε, την έκθεση που θέλαμε να υποβάλουμε. Επομένως, συμπερασματικά, με αυτή μας την εξέδεση μελέτες, καταλήξαμε στα ίδια, αλλά όλοι συμφωνούμε ότι λαμβάνουμε υπόψη τις απόψεις όσων ασχολήθηκαν και τα συμπεράσματα, τα επιστημονικά, θεωρήσαμε ότι δεν τεκμηριώνονται. Επίσης είναι σημαντικό το ότι δεν θα μπορούσαμε να ξάγαγουμε συμπεράσματα επί τη βάση αυτών των, των δειγμάτων που υπάρχουν των όσων έγιναν και κατόπιν της ανάλυσης που ακολούθησε. Και αυτό σε αυτό το άρθρο που δημοσιεύσατε είπατε ότι το δείγμα στο οποίο βασιστήκατε ήταν ε, πάρα πολύ μικρό σε σχέση με το να μπορούσαν να ληφθούν, ε, να αναξαχθούν κάποια αποτελέσματα σε σχέση με το αν υπάρχουν εδώ κάποια στοιχεία ε, τα οποία είναι τοξικά, τα οποία είναι, φέρνουν καρκίνο. Επομένω, δεν μπορούμε έτσι να θεωρήσουμε ότι για τον glyphosate έχουμε τεκμηριωμένη άποψη μέσω της μελέτης. Άρα, ακόμα περιμένουμε να, ξέρουμε κάποια άλλα συμπράσματα από κάποια έκθεση για τη μελέτη. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα αποτανθούμε στην Επιτροπή. Ο κύριος Λάντισλαβ Μίκο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα καταρχήν να καλωσορίσω τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης επανερχόμενο στη μελέτη του κυρίου Σεραλίνη μετά από τη ζωηρή συζήτηση πέρσι το φθινόπωρο και να σας μιλήσω για τη δράση μας έκτοτε. Καταρχήν θα ήθελα να τονίσω ότι η Επιτροπή κατέγραψε τη μελέτη και θεώρησε ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων έπρεπε να ασχοληθεί κατεπηγόντως με αυτήν. Ξέρετε τα συμπεράσματα της 28ης Νοεμβρίου του 12. Από τη δική μας άποψη θα ήθελα να τονίσω ότι η Επιτροπή δείχνει εμπιστοσύνη στα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια των ε, τροφίμων όλοι οι φορείς από τα κράτη-μέλη μπορούσαν να υποβάλουν ερωτήσεις εγκαίρως. Και θα ήθελα να τονίσω ότι έξι ε, τέτοιοι οργανισμοί κρατών μελών έφτασαν σε παρόμοια συμπεράσματα, τα οποία κατά την άποψή μου αποδεικνύουν την ασφάλεια της εργασίας της ΕΦΣΑ και την πληρότητα. Ο κύριος Σεραλίνη ε, έγειρε σοβαρά ζητήματα σε σχέση με τις ε, προαπαιτήσεις των, ε, στα κράτη-μέλη για την ασφάλεια των προϊόντων σε σχέση με τις μακροχρόνιες δοκιμές στους γενετικούς τροποποιημένους οργανισμούς και θα θέλαμε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανησυχίες. Είχαμε δύο εξελίξεις επί του θέματος. Πρώτον, η έγκριση του κανονισμού, τον προς ε, ε, έγκριση ε, ζωοτροφών και τροφίμων που περιέχουν γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Ο νέος κανονισμός επιβάλλει δοκιμές 90 ημερών για την τοξικότητα αναπερίπτωση και εάν υπάρχουν ενδείξεις αρνητικών επιπτώσεων θα πρέπει να διενεργηθούν διετής έρευνες. Η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη μιας μακροχρόνιας μελέτης για την τοξικότητα των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών, έτσι ώστε οι καταναλωτές να είναι σίγουροι για το υψηλό επίπεδο αποτίμησης κινδύνου αυτών των οργανισμών. Επίσης θα πρέπει σε ε, ορισμένες περιπτώσεις να γίνονται διετής ε, δοκιμές, ιδιαίτερα για ενδεχόμενες ε, καρκινογόνες ουσίες, κάτι το οποίο θα πρέπει να θεωρήσει ο κύριος Σεραλίνη ότι ισχύει. Ως προς την αυτονομία της ΕΦΣΑ, θα ήθελα να πω ότι η ΣΑΝΚΟ υποστηρίζει την ΕΦΣΑ, η οποία, ήδη, η οποία είναι αυτόνομη και αυτόβουλη και σύμφωνα με πρόσφατες ενδείξεις η ΕΦΣΑ και η ΕΜΑ είναι οι δύο πιο ε, αυτόνομοι κανονισμοί της, ε, οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να φτάσουμε σε κοινέ κατευθυντηρίες γραμμές για περίπτωση σύγκρουση συμφερόντων για όλους αυτούς τους οργανισμούς. Ως προς την πρόσβαση στα στοιχεία θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή στις 14 Ιανουαρίου έχει προβάλει μία πρωτοβουλία διαφάνειας για ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια στις εργασίες της αποτίμησης κινδύνων. Όλα τα στοιχεία θα πρέπει υπάρχουν για την παρουσία του NK603 ε, και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει, επειδή αυτά τα στοιχεία υπάρχουν στο διαδίκτυο, ε, θα πρέπει να μελετηθούν θεωρώντας ότι υπάρχει διαφάνεια επ' αυτών. Αυτή η πρωτοβουλία δεν αποτελεί αλλαγή της πολιτικής μας. Όλα τα επιστημονικά στοιχεία σε σχέση με τους γενετικούς, γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς έχουν αναφερθεί από την ΕΦΣΑ και δόθηκε θετική απάντηση στο NK603. Ως προς το glyphosate θεωρούμε ότι ε, ισχύει γι' αυτό ότι ίσχυε και για όλα τα άλλα φυτοφάρμακα από τις ε, εθνικές αρχές. Δηλαδή η Γερμανία έχει τα στοιχεία, υπάρχουν στη Γερμανία και εμείς δεν μπορούμε να διαδώσουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία κρατά στα χέρια της η Γερμανική Εθνική Αρχή. Επίσης, ως προς το glyphosate, θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να επανεκτιμήσουμε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για την ουσία glyphosate και πρόκειται για μία διαδικασία που άρχισε στη Γερμανία το Μάιο του 2012 και θα λήξει το Δεκέμβριο του 2013. Και επειδή η διαδικασία έγκρισης ισχύει μέχρι το 2015, αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις θα έχουμε μία πλήρη αποτίμηση των ε, πιθανών επιπτώσεων του glyphosate. Αυτό θα ήθελα να τονίσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ανοίγει η συζήτηση. Η κυρία Γκρέσε είναι η πρώτη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Πρώτα απ' όλα θέλω να χαιρετήσω το θάρρος και την επιμονή των αναφερομένων που ήρθαν εδώ και θέλω να τονίσω την υποστήριξη πολιτικής μου ομάδας προς αυτούς. Πριν από δύο μέρες, 25 Μαΐου, υπήρξε και μία διεθνής κινητοποίηση όπου εκατομμύρια πολιτών σε όλο τον κόσμο διαδήλωσαν κατά της Μονσάντο. Αυτό δείχνει ότι το θέμα το οποίο συζητούμε σήμερα απασχολεί όλους τους ανθρώπους στο πλανήτη μας. Θέλω να τονίσω ότι έχουμε πολύ μεγάλες αμφιβολίες για την αξιολόγηση κινδύνων με τους, σε σχέση με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Υπάρχουν πάρα πολλοί Πάρα πολλέ συγκρούσει συμφερόντων. Η κυρία Μπανάτη είναι πρόεδρος της ΕΑΤΕΦΣΑ και του ΣΕΑΤΙΝΣΕΡ, δηλαδή ενό οργανισμού ο οποίο χρηματοδοτείται από τι αγροτροφημικέ εταιρείε. Και επίση, θέλω να το τονίσω εξ ονομάτων ομάδα των Πρασίνων, είμαστε ιδιαίτερα ανίσχυοι σε σχέση με την αυξανόμενη επιρροή που ασκούν οι επιχειρήσει στα ερευνητικά θέματα, σε σχέση με τις καριέρες των επιστημόνων, σε σχέση με τις δημοσίευσεις. Και φυσικά υπάρχουν όλο και περισσότερες πιέσει για τις διαπραγματεύσεις που αφορούν εμπορικές συμφωνίες. Όλο και περισσότεροι πολιτικοί, όλο και περισσότεροι πολίτες ζητούν να υπάρξουν εγγύησεις. Δηλαδή να υπάρξουν πραγματικά επιστημονικές και ανεξάρτητες μελέτες κατά αντιπαράθεση και κατά αντιπολία και που να έχουν μακροχρόνιο χαρακτήρα. Θέλω να τονίσω εδώ ότι θα υπάρξει εμπιστοσύνη στην ΕΦΣΑ μόνο όταν εξαλειφθούν οι συγκρούσει συμφερόντων σε όλα τα επιστημονικά πάνελ, σε όλα τα δικηδικά όργανα τη ΕΦΣΑ. Και φυσικά έχω πάρα πολλά ερωτήματα. Μερικά από αυτά τα ερωτήματα. Μήπω θα πρέπει να ξανασκεφτούμε τι διαδικασίε επιστημονική εμπειρογνωμονησύνη τη ΕΦΣΑ. Μήπω η ΕΦΣΑ θα πρέπει να επανεξετάσει τη μεθοδολογία της για την αξιολόγηση των κινδύνων. Γιατί η ΕΦΣΑ έχει αρνηθεί να γίνουν μακροχρόνιες τοξικολογικές μελέτες. Και προς την Κομισιόν τώρα. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ να ξέρω τι κάνει η Κομισιόν για να υποστηρίξει την ΕΦΣΑ στον ρόλο της που είναι υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, ώστε εν τέλει οι πολιτικοί και οι άνθρωποι στην Ευρώπη να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ανεξάρτητες μελέτες. Και επίσης επειδή είμαστε πολλοί οι βουλευτές από όλες τις πολιτικές παρατάξεις που στείλαμε μια επιστολή προς την Κομισιόν για το θέμα αυτό και προτείναμε να υπάρξει και ένα νομοθετικό πλαίσιο για τα θέματα των διαδικασιών εμπειρογνωμοσύνης και αντιμετώπισης συγκρούσεως συμφερόντων. Ποια είναι η κατάσταση στην Κομισιόν αυτή τη στιγμή. Και τέλος, η ομάδα των Πρασίνων έχει την θέση που πιστεύω ότι υποστηρίζεται από τους περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες όταν, όπως φάνηκε και από τις δημοσκοπήσεις. Όσο υπάρχουν κίνδυνοι, όσο υπάρχουν αμφιβολίες, υπάρχει η απόλυτη ανάγκη να υπάρξει ένα μορατόριο για οποιαδήποτε χρήση καλλιεργειών γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρος. Έχετε το λόγο κύριε Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους αναφερόμενους γιατί μας ε, εφιστούν την προσοχή σε ένα βασικό πρόβλημα και εδώ οι νομοθέτες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν θεσπίσει ένα φορέα την ΕΦΣΑ που είναι αρμόδιος για τα θέματα αυτά. Οι αναφερόμενοι θέλουν να εξασφαλίσουν την ανεξαρτησία της ΕΦΣΑ. Εμείς ως Επιτροπή Αναφορών αντιμετωπίζουμε εδώ δυσκολίες γιατί πρόκειται για ορισμένα προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα. Η ζωή περιλαμβάνει και τους κινδύνους. Όταν μιλάμε για μηδενικό κίνδυνο, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρξει ζωή χωρίς κίνδυνο. Και το θέμα είναι βέβαια πώς ταξινομούμε τους κινδύνους και πώς τους ιεραρχούμε. Ένα φιλοσοφικό θέμα, αλλά περιμένουμε από μια αρχή όπως η ΕΦΣΑ να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία των εργασιών τους. Τι είναι όμως τώρα πραγματικά ανεξάρτητο. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος ο οποίος είναι απόλυτα ανεξάρτητος και απόλυτα χωρίς να έχει κάποιες συνδέσεις και κάποια συμφέροντα. Μια τρίτη παρατήρηση. Η ΕΦΣΑ προσπαθεί να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της, αλλά πρέπει συγχρόνως να εξασφαλίσει και την πραγματική εμπειρογνωμοσύνη. Πώς λοιπόν εξασφαλίσουμε την εξισορρόπηση μεταξύ της ανεξαρτησίας και της γνώσης, της ε, εμπειρογνωμοσύνης. Εάν λοιπόν θέλουμε ε, ε, ανεξαρτησία, αλλά αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι καταλαβαίνουν κάτι για το επιστημονικό υπόβαθρο θεωρούνται λομπίστες και οι μόνοι οι οποίοι θεωρούνται ανεξάρτητοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα, τότε αυτό δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε θετικά συμπεράσματα. Εγώ ως μέλος της Επιτροπής της ε, Επιτροπής Αναφορών δεν θεωρώ ότι είμαι σε θέση να λύσω αυτό το κουβάρι, γιατί εδώ πρέπει τα θέματα αυτά να τα αντιμετωπίσουν οι εμπειρογνώμονες. Θέλουμε να τα συζητήσουν τα θέματα αυτά οι εμπειρογνώμονες, θέλουμε η ΕΦΣΑ να μπορέσει να αποφασίσει με έναν τρόπο ο οποίος είναι ανεξάρτητος και αμερόληπτος. Αλλά εγώ φοβάμαι ότι όποιο θεσμό και να πάρει κανείς για να εξετάσει πάντα μπορεί να προκύψει μια συζήτηση για την ανεξαρτησία του θεσμού αυτού. Και εγώ νομίζω ότι τα θέματα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουν οι εμπειρογνώμονες και οι ειδήμονες στα θέματα αυτά. Εγώ δεν θέλω να πω ότι δεν υπάρχει λόγος για μια υποψία σε αυτήν την περίπτωση, αλλά εγώ πραγματικά θεωρώ ότι σαν μέλος της Επιτροπής Αναφορών δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τα επιστημονικά και νομικά θέματα τα οποία συνάπτονται με αυτήν την ε, αναφορά. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Επιτροπή μας να παραπέμψει αυτό το θέμα σε άλλες επιτροπές, γιατί δεν νομίζω ότι εμείς μπορούμε να βρούμε την άκρη του κουβαριού. Έχω μία μόρφωση, δεν ε, μπορώ να θεωρήσω ότι και εγώ ο ίδιος είμαι απόλυτα ανεξάρτητος, αλλά πραγματικά το ερώτημα τι θα πει ανεξαρτησία και ποια είναι τα όρια της ανεξαρτησίας. Εμείς θα πρέπει λοιπόν να λειτουργήσουμε και να παίξουμε το ρόλο μας και δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει απόλυτη ανεξαρτησία κανός, κανός φορέα. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει η καταγραφή των προβλημάτων. Το θέμα είναι να βρούμε και μια λύση η οποία θα είναι ουσιαστική. Και αυτό είναι ένα θέμα για τους εμπειρογνώμονες. Εγώ χαίρομαι που υπάρχει ΕΦΣΑ, θα πρέπει να αποφασίσει και πάντα αυτός ο οποίος παίρνει απόφαση, αυτός είναι αυτός ο οποίος ε, υπόκειται και σε κριτική. Και ακριβώ αυτό σημαίνει και ανεξαρτησία. Να μπορεί κανεί να παίρνει αποφάσει οι οποίε θα τη χάνουν επικρίσεων. Κύριο Τέιλορ. Yes, thank you very Ευχαριστώ πολύ. να ευχαριστήσουμε τον αναφέρομενο που ήρθε εδώ Ευχαριστούμε ότι ο ίδιο. Ελπίζουμε ότι ο ίδιο μπορεί να δώσει απαντήσει όσον αφορά την προσβασιμότητα ε, στην ε, έκθεση, τη μελέτη αυτή, γιατί εμένα ε, θα με εξέλιξε πάρα πολύ το να μην μπορούσε η ΕΦΣΑ να έχει πρόσβαση στην μελέτη του κύριου Σελήνη. Γιατί χρειαζόμαστε και τη δική σας μελέτη. Αυτή τη στιγμή ακριβώ πούμε, με τι κλινικέ δοκιμέ, τα κλινικά πειράματα. Και ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει με επιτυχία και θα μπορούμε να έχουμε πλήρη διαφάνεια. Για αυτά τα πρωτογενή δεδομένα ακριβώ όπω είπατε στην αρχή. Και ελπίζουμε να συνεχίσει να είναι μερόληπτο ο διαμεσολαβητή όπω είναι τώρα. Κλασικά έτσι είναι. Ακριβώ όπω επεφάνθη πριν από δύο χρόνια να να που αφορούσε την αίμα ε, Ήταν η υπόθεση 1049 για την διαφάνεια και ξεκαθάρα είχε κρίνει ότι όταν έπεσε την αίμα θα πρέπει να ε, αποκαλύψει, να δημοσιεύσει την μελέτη, τότε Και εμείς θελήσαμε ότι θα πρέπει τα πρωτογενή στοιχεία να είναι προσβάσιμα. Αυτά όλα στα οποία στηρίχθηκε η έγκριση για να χρησιμοποιούνται αυτές οι ουσίες. Δηλαδή να είναι δυνατόν όλοι, όλοι να έχουν πρόσβαση, γιατί αυτό αφορά τους πολίτες. Και έχουμε και τη σύμβαση του όρχους, Εκτό από την απόφαση του Διαμεσολαβητή. Μα είναι τόσο δύσκολο να τα καταλάβει αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω η ΕΦΣΑ τουλάχιστον το κατάλαβε ότι χρειάζεται να υπάρχει διαφάνεια και να μπορεί στα προγενή δεδομένα να έχει πρόσβαση ο κόσμο. Και εσείς βέβαια, κύριε καθηγητά, θα πρέπει να δίνετε τα δεδομένα σας. Τα στοιχεία σας. Κύριε Γιάρ, υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν θεσπιστεί ε, στο διοικητικό δίκαιο της κάθε χώρας, οπότε θα πρέπει αυτά να ισχύουν και σε ενωσιακό επίπεδο, γιατί σύμφωνα με την συνθήκη, την σχετική, υπάρχει το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση, οπότε και εκεί υπάρχουν αντικειμενικά πολύ συγκεκριμένα κριτήρια σε σχέση με τα προσωπικά ή τα οικονομικά κριτήρια. Ας πούμε, κάποια νου να δουλεύει ε, εν λόγω η εταιρεία, η σύζυγος. Δηλαδή, όσο και κανείς δεν είναι νομοταγής, θα πρέπει να εξετάζεται αν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων. Άπαξ και διακυβεύονται κάποια προσωπικά του συμφέροντα λοιπόν ή κάποια χρήματα. Ε, Βεβαίω και θα πρέπει όλου να του εξετάζουμε αν έχουν σύγκρουση συμφέροντα, γιατί πρόκειται να μιλάμε για μισό εκατομμύριο ανθρώπους στην Ευρώπη. Μισό δισεκατομμύριο. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μετά από αυτά που λέει η Μάργαρετ δεν μπορώ να πω πολλά. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι πράγματι τα θέματα της σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε περισσότερο. Όλοι θέλουμε ανεξάρτητες μελέτες αλλά κυρίως θέλουμε την πρόσβαση στα στοιχεία. Γιατί έχουμε δει πόσο μπερδεμένα είναι τα πράγματα με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και πόσο μεγάλη αντιπαράθεση υπάρχει για τα θέματα αυτά. Εγώ νομίζω ότι ακόμα και οι μαθητές του γυμνασίου καταλαβαίνουν ποια είναι τα θέματα της ε, τοξικότητας και τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν. Το ήταν και αντικείμενο συζήτηση σε ένα σχολείο στην εκλογική μου περιφέρεια και θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον αναφερόμενο για το θάρρος του. Κυρία Σεραλίνη, θέλετε να λάβετε το λόγο. Πολύ σύντομα. Καταρχήν, Για άλλη μια φορά θα ήθελα να πω ότι το γλυφοσάτ και διακόπτει ο μιλητής. Σας παρακαλώ εντάχει. Εγώ είχα ζητήσει το λόγο και σας ευχαριστώ που μου τον δίνετε, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη, κύριε καθηγητά. Ήθελα να παρέμβω σε αυτό το σημαντικό ζήτημα ευχαριστώντας τους αναφέροντες γιατί πραγματικά επέμειναν και πολύ σωστά. Και να ευχαριστήσω και τον ε, καθηγητή Σεραλίνη για την παρουσία και την ε, παρέμβασή του. Έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα όπου υπάρχουν πολύ μεγάλα συμφέροντα. Στον ιδιωτικό, επιχειρηματικό τομέα, καθώς και από τον δημόσιο θέματα κοινωνικού συμφέροντος και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό και υπάρχουν και μεγάλες δυσκολίες αντιμετώπισης του θέματος. Θα ήθελα να ρωτήσω τον καθηγητή Σεραλίνη, εάν μπορεί να μας ε, διευκρινίσει κάπως το εξής, γιατί η μελέτη του είχε εμπιστευτικό χαρακτήρα για μια μεγάλη χρονική περίοδο, δηλαδή κατά τη διενέργεια της μελέτης. Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισε ο καθηγητής κατά τη διενέργεια της έρευνας και ποιοι ήταν οι οικονομικοί η χρηματικη υποστήριξη που έλαβε για την εκπλήρωση αυτής της εργασίας. Και όταν ολοκληρώθηκε αυτή η έρευνα, οπωσδήποτε είχε μία πολύ μεγάλη απήχηση. Και είχε αυτή την εμβέλεια διότι είναι ένα ζήτημα ύψης της σημασίας, μιλάμε για πρόσβαση στα στοιχεία, για τη διαφάνεια, για θέματα διαφάνειας, γιατί έχουμε να κάνουμε με μικρές ομάδες ερευνητών και ε, επιστημονικές δυνάμεις που δίνει τιτάνιο αγώνα κατά των μεγάλων ε, επιχειρήσεων. Η Μονσάντο είναι μία από αυτές που έχει μεγάλη, μεγάλες οικονομικές δυνατότητες καθώς και δυνατότητα επιρροής. Καταλαβαίνουμε ότι σε όλες τις υπήρους υπάρχουν καταστάσεις ε, σύραξης, θα μπορούσα να πω διαφοράς, διαφορών μεταξύ της Μονσάντο και επιστημονικών κοινοτήτων, αγροτών, εκτροφέων που δεν δέχονται τη δραστηριότητα της ε, Μονσάντο και αυτό το καταδεικνύει και η έρευνα αυτή. Είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι μπροστά σε αυτή την κατάσταση και θεωρούμε ότι η αρχή της πρόληψης είναι ύψη της σημασίας. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να δέχονται τρόφιμα που εμπεριέχουν γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς η επίπτωση των οποίων δεν είναι απόλυτα γνωστή. Αυτό το ξεχνάμε όλο ένα και περισσότερο και δεν λαμβάνεται τόσο σοβαρά υπόψη. Και εδώ ε, ανακύπτουν ακριβώς οι κίνδυνοι για τον πληθυσμό και γι' αυτό υπάρχουν και μεγάλες διαμαρτυρίες προβάλλονται όλο ένα και περισσότερες διαμαρτυρίες εναντί αυτών των ε, κινδύνων. Επίσης, έχω την εντύπωση ότι η Επιτροπή κρατά αμυντική στάση και αυτό έχει γίνει ήδη εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Δηλαδή, θεωρεί ότι οι χώρες αυτές ήδη έχουν τιμιγορήσει. Μιλάμε για τις έξι αυτές χώρες και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να τις δούμε ως μια μειοψηφία τις έξι χώρες δηλαδή έναντι των 27 που είναι πιο οργανωμένες. Νομίζω λοιπόν ότι ε, δεν θα πρέπει να υπάρξει αυτή η θεώρηση του ζητήματος. Τώρα θα πρέπει να μας πει η Επιτροπή κατά πόσο θα διενεργηθούν περαιτέρω έρευνες και μελέτες το 2013. Ίσως θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί και εκ των προτέρων. Και ως προς τη, ε, το κατά πόσο αυτοί οι οργανισμοί είναι ανεξάρτητες αρχές, θα πρέπει να δούμε το θέμα ε, κατά αντιπαραβολή ιδιωτικών και δημοσίων συμφερόντων. Σε κάθε χώρα ε, υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση όμως, εν κατακλείδη, μπορούμε να πούμε το εξής. Τη στιγμή που οι δημόσιοι φορείς και ερευνητικά κέντρα καταργούνται και τα ερευνητικά κέντρα προωθούνται μόνο στα πλαίσια των μεγάλων επιχειρήσεων, δηλαδή του ιδιωτικού τομέα, καταλαβαίνουμε ποια είναι η πραγματική ε, αυτονομία αυτών των ερευνητικών οργανισμών. Γιατί η ζωή τους εξαρτάται από την ιδιωτική επιχείρηση. Αυτό είναι σαφές. αυτό το ζήτημα, αυτή η διάσταση του ζητήματος μας ε, δείχνει ότι θα πρέπει να βασιστούμε σε δημόσιους οργανισμούς, σε ερευνητικούς οργανισμούς που πραγματικά είναι αυτόνομοι και αυτόβουλοι, όπως προαπαιτείται. Άρα, θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να ακολουθήσουμε την αρχή της ε, πρόληψης έτσι ώστε να μην φτάνουν στον καταναλωτή προϊόντα που δεν είναι ασφαλή. Που, για το οποίο δεν ξέρουμε αν πραγματικά είναι τοξικά ή όχι. Και αυτό αφορά και τις ε, ζωοτροφές. Δεν πρέπει να γίνεται αδιάκριτη χρήση ορισμένων ουσιών που μακροχρόνια θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο ή αντίθετο από αυτό που προβάλλεται βράχη πρόθεσμα. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε. Ο καθηγητής Σεραλίνη έχει το λόγο και πάλι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος για κάθε σημείο. Κύριε Επίτροπε, εκπρόσωπε της Κομισιόν καλύτερα. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το glyphosate δεν ταυτίζεται με το Roundup. Το Roundup περιλαμβάνει πάρα πολλές χημικές ενώσεις, κάποιες από τις οποίες είναι πιο τοξικές για τα θηλαστικά και τον άνθρωπο από ότι το glyphosate. Και κανείς, κανένας φορέας που αναφέρατε αντιμετωπίζει την μακροχρόνια αξιολόγηση του Roundup. Και το Roundup είναι το μεγαλύτερο παρασιτοκτόνο στον κόσμο 80% των βρόσιμων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών έχουν δημιουργηθεί για να απορροφούν το Roundup. Ελπίζω ότι είμαι σαφές, σαφής στο θέμα αυτό. Μέχρι σήμερα η ΕΦΣΑ δεν μπορεί να δώσει τα πρωτογενή, τα κατέργαστα στοιχεία, όχι μονάχα για το γκλαϊφοσάτ, αλλά και για τα πάρα πολύ σύντομου ορίζοντα τεστ που έχουν γίνει από τα κράτη-μέλη λιγότερα από 10 ζώα για το Roundup και για τους ερθισμούς στα μάτια και στο δέρμα που προκαλεί. Αυτό είναι ένα πραγματικό υγειονομικό πρόβλημα. Έχετε 150.000 προϊόντα και κάποιες χιλιάδες παραστοκτόνων που αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Εγώ συμφωνώ ότι η ΕΦΣΑ και άλλοι φορείς πρέπει να είναι υπεύθυνε για την αξιολόγηση των προϊόντων, αλλά δεν έχουν τον εξοπλισμό, δεν έχουν τον εξοπλισμό για να το κάνουν αυτό. Και έχουν προβλήματα σύγκρουση συμφερόντων. Υπάρχει τεράστιο οικονομικό συμφέρον που συνδέεται με τα θέματα αυτά. Εδώ και 20 χρόνια όλα τα κράτη-μέλη έχουν ζητήσει από τα πανεπιστήμια τους να συνεργάζονται με τη βιομηχανία. Υπάρχει μια συντεχνιακή λοιπόν σχέση που έχει οδηγήσει σε ορισμένες παγιωμένες πρακτικές, όπως χάρη η χρήση των ιστορικών στοιχείων. Επίση, υπάρχουν συγκεκριμένες συνδέσεις συμφερόντων. Η πρότασή μας προς την ΕΦΣΑ είναι και οι δύο πλευρές να δώσουμε στη δημοσιότητα τα πρωτογενή μας στοιχεία. Ήρθαμε τότε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάναμε μια ανακοίνωση τύπου και είπαμε ότι είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα στοιχεία μας, να δοθούν όλα στο διαδίκτυο και όχι μονάχα στην ΕΦΣΑ και θα το κάνουμε αυτό με την προϋπόθεση ότι θα το κάνει και η ΕΦΣΑ και ζητήσαμε να δοθούν στη δημοσιότητα όλα αυτά τα στοιχεία και θα ήθελα να γίνεται αυτό όχι μόνο για το Roundup αλλά και για όλα τα προϊόντα που έχουν να κάνουν με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Είναι απαραίτητο να υπάρχει αυτή η διαφάνεια λοιπόν. Δεν θέλω να δαπανηθούν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν εξασφαλίσουμε πρώτα αυτή τη διαφάνεια. Γιατί δεν θα μπορούμε να ερμηνεύσουμε σωστά τα πρωτογενή στοιχεία οποιασδήποτε μελέτης. Και πάλι εδώ υπάρχει ένας συμβολικός λόγος για τον οποίο εμεί δεν δώσαμε στην ΕΦΣΑ τα στοιχεία αυτά, αλλά μόνο στο περιοδικό Food and Chemical Toxicology και σε άλλους επιστήμονες. Ο Ρίτσαρντ Γκούτμαν, ο συντάκτης της Biotech, πέρασε, ε, ε, ζήτησε από την Food and Chemical Toxicology να ερευνήσει ορισμένα ε, άρθρα και το περιοδικό αυτό ε, αφήρεσε ένα άρθρο που είχε δεχτεί στο παρελθόν. Και επίσης ο, ο, αρχισυντάκτης του Transgenic Research όταν το ρώτησα τι είναι είπε ότι υπάρχουν προβλήματα με ψευδοεπιστημονικά άρθρα και είπε ότι η δημοσίευση του δικού μου άρθρου ήταν ένα λάθος. Αλλά υπάρχει σύνδεση γιατί υπάρχουν ε, ευρεσιτεχνίες μεταξύ αυτών οι οποίοι ασχολούνται με τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Και συμφωνώ ότι θα πρέπει να είναι ενδιαφέρον να βρούμε πώς θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο δεν έχει ε, συγκρούσεις συμφερόντων. Γι' αυτό ζητούμε από την Κομισιόν και από το Συμβούλιο των Υπουργών να υπάρξει δυνατότητα κατά αντιμολία, κατά αντιπαράθεση εμπειρογνωμοσύνης με στόχο να καταλήξουμε σε μία ανεξάρτητη γνώμη και όχι μόνο να υπάρξει αντιπαράθεση απόψεων, αλλά πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια για τα πρωτογενή στοιχεία. Όχι λοιπόν μονάχα να προσπαθούμε να βρούμε ανεξαρτησία μέσα εισαγωγικά στα πανεπιστήμια που είναι όλο και πιο εξαρτημένα από τη βιομηχανία γιατί χρηματοδοτούνται από τη βιομηχανία αντί να ακολουθούμε αυτό το δρόμο θα πρέπει να ζητήσουμε κάτι που κοστίζει 0 ευρώ και αυτό δεν είναι θέμα της ΕΦΣΑ θα πρέπει να ζητήσουμε να υπάρχει διαφάνεια σε σχέση με τα πρωτογενή στοιχεία. Εάν συμφωνήσει η Κομισιόν, αυτό μπορεί να υλοποιηθεί αύριο. Και με την διαφάνεια αυτή μπορούμε να έχουμε τα στοιχεία αυτά και για τις αιματολογικές μελέτες. Γιατί αυτή τη στιγμή το Roundup είναι μυστικό σε σχέση με την ε, σύνθεσή του, επομένως δεν μπορούν να γίνουν οι τοξικολογικές μελέτες και γι' αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια ανάλυση. Και θα ήθελα να κλείσω λέγοντας γιατί το θέμα αυτό δεν έχει φτάσει ένα ευρύτερο κοινό. Στην Φιγαρό, ο Ζεράρ Πασκάλ έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι αυτό το άρθρο δεν είναι σωστό. Χρειάστηκαν τέσσερις μήνες για να το δημοσίευσει το περιοδικό στο οποίο δημοσιεύτηκε και μέσα σε μία μέρα οι εφημερίδες είπαν ότι αυτό το άρθρο δεν σημαίνει τίποτα και δεν ήξεραν ότι το άτομο το οποίο έδωσε την συνέντευξη ήταν αυτό που κατάφερε να αποφύγει να γίνουν μελέτες πέραν των τριών ε, μηνών για το NK603. Και επίσης αυτός έχει συμμετάσχει στο διορισμό, διαδικασία διορισμού των εμπειρογνωμόνων στο, στην ΕΦΣΑ και επίσης συμμετέχει σε ένα υποτίθεται ανεξάρτητο οργανισμό αξιολόγησης στη Γαλλία. Υπάρχουν πάρα πολλές λοιπόν συγκρούσεις συμφερόντων οι οποίες δεν αποκαλύπτονται. Τις ξέρω συγκεκριμένα και ονομαστικά γιατί εγώ είμαι σε αυτό το γκεζί, είμαι σε αυτή τη διαδικασία. Πριν από 9 χρόνια ήμουν εκεί και βγήκα από αυτή για να μπορέσω να κάνω αυτό το πείραμα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Λίγη αυτή η εισβάθο συζήτηση με μεγάλες συμμετοχές. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα διαφάνειας, ουσιώδους διαφάνειας και συμμετοχής ακόμα και των πολιτών μαζί με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Πολλοί συνάδελφοι κατά την παρέμβασή τους ζήτησαν από την Εύσα να κοινοποιήσει τα στοιχεία, τα λείποντα στοιχεία, που να ε, επιτρέπουν στους πολίτες άμεση πρόσβαση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να προωθηθεί έτσι ώστε να μας απασχολήσει περαιτέρω. Πέρα από αυτό το θέμα της διαφάνειας, και της αρμοδιότητας, της ε, θεσμικής αρμοδιότητας με την τροποποίηση των ε, ευρωπαϊκών κανονισμών ίσως θα πρέπει ε, να ζητήσουμε γνωμοδότηση από τις καθήλυν αρμόδιες επιτροπές, όπως είπε και η συνάδελφος Γιάρ. Αναφέρομαι στην Επιτροπή, στις Επιτροπές Γεωργίας και Περιβάλλοντος που ίσως επί της ουσίας θα μπορούσαν να μας υποστηρίξουν. Θα ήθελα όμως αυτό το θέμα, αυτή την αναφορά να την αφήσουμε ανοιχτή έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, καταγράψουμε και τα όσα ε, προανέφερε, όσα, σε όσα αναφέρθηκε ο αναφέρον δηλαδή να καταγράψουμε τις σημειώσεις του. Θα γίνουν περαιτέρω διερευνήσεις και παραμένει το αίτημα προς την ΕΦΣΑ για μεγαλύτερη διαφάνεια και η Επιτροπή να μας δώσει περισσότερες διευκρινήσεις. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες, ιδιαίτερα τον καθηγητή Σεραλίνη και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων και προς το επόμενο θέμα την αναφορά της κυρίας ε, Βίκε Ράινχαρτ, γερμανικής ηθαγένειας. Η αναφορά συνοδεύεται από 2.500 υπογραφές σε σχέση με την ομοιόμορφη σήμανση των γενετικά τροποποιημένων ζωοτροφών και τροφίμων. Από κοινού θα μας απασχολήσει η αναφορά 807 κάθετος 2012 του Μισελ Γκροσχάρτ. Οι αναφέροντες δεν είναι παρόντες, γι' αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Λάτεσλαβ Μίκο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα με γρηγορήσω όσον αφορά την σήμανση. Σας επαναλαμβάνω ότι είναι πάρα πολύ ύψιστη η προτεραιότητά μας γιατί θέλουμε να υπάρχει ασφαλεία σε σχέση με τους συγκεκριμένους τροποποιημένους ε, οργανισμούς. Και όσον αφορά αυτή την σήμανση, δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε με τον Ετούντα τι Είναι ετούσα τελεσοδετωμένη σε σχέση με το ότι θέλει να υπάρχει ομοιόμορφη σήμανση και έτσι να μπορεί να κατοχυρωθεί η ελεύθερη επιλογή. Επίσης, σας ε, θυμίζω ότι στην Ευρώπη ισχύει σχετική νομοθεσία. Ε, αναφέρεται εδώ επομένω ότι ε, κάποιες, ε, κάποιοι τέτοιοι οργανισμοί δεν έχουν τύχει εγκρίσεως και είναι παρόντες σε αυγά γαλακτοκομικά ή κρέα. Παρ' όλα αυτά δεν αποκλείει νομοθεσία το να υπάρχουν κάποιες, ε, υπάρχει κάποια σήμανση που να μην αναφέρει τους, τους οργανισμού οργανισμούς που υπάρχουν στο τρόφιμο. Κάναμε εμείς μια μελέτη όσον αφορά το βεληνικές αυτών των ετικετών αυτής της ε, επισήμανσης και είπαμε ότι θα πρέπει να προχωρήσει η εναρμόνιση θα υπάρξει μια μελέτη και θα δημοσιευθεί περί τα μέσα του έτους. Συμφωνώ με τους ετουμένους ότι δεν θα πρέπει ε, αυτές οι ζωοτροφές να μην ανακατεύονται με, με γενετικά τροποποιημένα. Οπότε κατακλείδη είναι δικαίωμα του καταναλωτή να υπάρχει τέτοια πλήρης ε, σήμανση και πλήρης ε, ενημέρωση του καταναλωτή και γι' αυτό και θέλουμε να υπάρξει ε, ε, σήμανση με τέτοια που να λέει αν, αν απουσιάζουν και να περιμένουμε να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες από ό,τι σήμερα. Ο κύριος Χιάρ Συμφωνούμε όλοι κύριε Πρόεδρε. ότι είναι ανθρώπινο δικαίωμα να ξέρει κανείς τι είναι αυτό που αγοράζει και πώς παράγονται τα προϊόντα αυτά. Και αυτό ισχύει πολλό μάλλον για τα τρόφιμα. Είναι θέμα βασικής διαφάνειας να ξέρουμε τι είναι αυτά τα οποία τρώμε. Και για την ε, γενετική μηχανική πολλές φορές είναι πολύ λίγα τα πράγματα τα οποία γνωρίζουμε. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό ισχύει όχι μόνο για τα τρόφιμα, αλλά έχει να κάνει και με τα φάρμακα τα οποία ε, παίρνουμε όλοι μας. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε αν έχει χρησιμοποιηθεί γενετική μηχανική ή όχι στην παραγωγή τους. Πολλοί δεν ξέρουν ότι τα περισσότερα ε, τυριά παραγόνται με μια διαδικασία ζύμωσης η οποία δημιουργεί γενετικές τροποποίησεις. Και πολλές φορές λέμε ότι για να το ξέρει, για να το ξέρει αν έχουν ε, γενετικά τροποποιημένα προϊόντα πρέπει να γυρίσουμε πίσω και να φτάσουμε ως την Αγελάδα και να ξέρουμε τι ακριβώς έχει φάει η Αγελάδα και αν είναι τροποποιημένο ή όχι. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η πρόθεση και η διαδικασία να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια γιατί πάρα πολλοί πολίτες θέλουν να έχουν μεγαλύτερη διαφάνεια για το από πού προέρχονται τα, τα προϊόντα που καταναλώνουν και αυτό φάνηκε και από την προηγούμενη συζήτηση. Πρόκειται για μια νέα τεχνολογία λοιπόν. Χρειάζεται αυτή η τεχνολογία περαιτέρω έρευνα για τα θέματα αυτά και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει τι απαραίτητε μελέτε και δεν κάνει την αξιολόγηση του κινδύνου, τότε θα τα κάνουν πολλοί άλλοι. Και ένα μεγάλο μέρο από την έρευνα για του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού δεν γίνεται πια στην Ευρώπη. Έχει ξεφύγει από την Ευρώπη. Αν δεν τα κάνουμε λοιπόν εμείς αυτά, δεν κάνουμε την απαραίτητη έρευνα και αξιολόγηση κινδύνου, τότε το κάνουν τρίτη για μας. Τέλος. Εγώ υποστηρίζω απόλυτα την ε, πλήρη διαφάνεια να ξέρουν όλοι αυτοί οι καταναλωτές τι τρώνε, τι, αφορού, τι καταναλώνουν, αλλά πρέπει να ισχύει όχι μόνο για τη λεγόμενη πράσινη βιοτεχνολογία, αλλά και για τη λεγόμενη κόκκινη και άσπρη βιοτεχνολογία για όλες τις ε, διαδικασίες που χρησιμοποιούν τέτοιες τεχνολογίες. Γι' αυτό πιστεύω πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή την ε, ε, αναφορά αυτή και να περιμένουμε τα αποτελέσματα των μελετών για τα θέματα αυτά. Κάποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο. Όχι. Ναι, ναι, παρακαλώ. Ο Τσικόφσκι. Συγγνώμη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής. Αλλά λόγω του περιεχομένου αυτών των ε, αναφορών ήρθα εδώ. Χαίρομαι που έχει εξεταστεί αυτή η αναφορά και εγώ υποστηρίζω απόλυτα την ιδέα ότι όλα τα προϊόντα που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς θα πρέπει να την χάνουν ιδιαίτερη σήμανση για να διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα προϊόντα. Συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Γιάρ και μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την έρευνα να συμμετέχουν όχι μόνο άτομα που είναι εμπειρογνώμονες στη βιοτεχνολογία, αλλά να υπάρχουν και ερευνητές οι οποίοι εξετάζουν την επίπτωση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην ανθρώπινη και ζωική υγεία και στο περιβάλλον. Εκεί πρέπει να είναι το αποφασιστικό στοιχείο. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε τους ίδιους ανθρώπους που έχουν συμφέρον σε μια διαδικασία να κρίνουν τον εαυτό τους. Ο σημαντικός ρόλος θα πρέπει να είναι λοιπόν ο έλεγχος του αντίκτυπου στην ανθρώπινη υγεία. Σας ευχαριστώ. Καλώς ήλθατε στην Επιτροπή Αναφορών. Αν δεν υπάρχει λοιπόν κάποιος συνάδελφος, μπορώ να πω ότι είναι σαφές ότι οι παρεμβάσεις ζήτησαν να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και θα παραμείνει επομένω ανοιχτή. Πάμε στην, στο σημείο 7 για την ε, αναφορά που έχει να κάνει με δύο αιωλικά πάρκα που έχουν εγκατασταθεί στην μεθοριακή περιοχή του Ού στην και αφορά τον αντίκτυπό τους στις ε, όμορες ε, περιοχές της Γερμανίας. Ο κ. Σόκμα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμμετείχα σε αυτή τη συζήτηση αυτής της Επιτροπής ε, αρκετές φορές. Θα ήθελα λοιπόν να συνοψίσω τις πρόσφατες εξελίξεις από το Φεβρουάριο όταν αρχικά συζητήθηκε αυτό το ζήτημα. Οι τσεχικές αρχές περιβάλλοντος μετά από διενέργεια έρευνας για τον αντίκτυπο επί του περιβάλλοντος έφτασαν σε ένα συμπέρασμα τον Απρίλιο το αποτέλεσμα κοινοποιήθηκε στις γερμανικές αρχές τον Απρίλιο, νομίζω στις 19 Απριλίου και οι τσεχικές περιβαλλοντικές αρχές δημοσίευσαν στα τσεχικά και στα γερμανικά τα συμπεράσματα της δημόσιας ιστοσελίδας του Οργανισμού Περιβάλλοντος. Η Επιτροπή ε, εξέτασε εκ του σύνεγγης αυτή τη διαδικασία και από πλευράς ε, διαδικαστικής καθαρά δεν βλέπουμε καμία παραβίαση των προδιαγραφών. Επί της ουσίας, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αποφασίσει κατά πόσο υπάρχει κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει εκ νέου. Στο μεταξύ όμως ε, λάβαμε ε, μία προσφυγή που, η οποία ε, πρωτοκολλήθηκε αυτό το μήνα. Με βάση αυτό το αίτημα θα δούμε κατά πόσο θα πρέπει να φυγεί αυτό το ζήτημα με τις τσεχικές αρχές. Προς το παρόν, η Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο, διότι δεν μπορεί να εκινήσει μία διαδικασία επί παραβάση για ένα θέμα το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν ακόμα ε, ε, ε, πρόκειται για μια εκρεμή διαδικασία, γι' αυτό ακόμα δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Γιάρ. Ο κύριος Γιάρ. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, αυτά τα σχέδια για ένα αιωλικό πάρκο κοντά στα γερμανικά σύνορα. Πρόκειται για τουρμπίνες που θα φτάνουν τα 150 μέτρα και βρίσκονται δίπλα σε ένα χώρο ο οποίος την χάνει οικολογικής προστασίας. Πρέπει λοιπόν η Επιτροπή η οποία κάνει την ε, αξιολόγηση αυτού του σχεδίου να αντιμετωπίσει και τις μεθοριακές, διαμεθοριακές συνέπειες οι οποίες θα προκύψουν και στη γειτονική χώρα, δηλαδή στη Γερμανία. Να υπάρξει λοιπόν η... να υπάρξει και συμμετοχή από τους αρμόδιους της άλλης πλευράς. Και γι' αυτό έχω διατυπώσει την πρόταση και οι δύο χώρες από κοινού να προβούν σε αυτή την αξιολόγηση. Όταν λοιπόν πρόκειται για τέτοιου είδους σχέδια τα οποία βρίσκονται σε μεθοριακές περιοχές που υπάρχει κάποια επίπτωση και τις δύο πλευρές είναι απαραίτητο να υπάρχει μια κοινή αξιολόγηση. Αυτό απορρέει και από την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο συγκεκριμένο στοιχείο, εδώ η Κομισιόν μας είπε ότι υπάρχει αυτή, αυτό το παράπονο. Εδώ το ερώτημα που θέλω να θέσω είναι το εξής. Θεωρεί η Κομισιόν ότι πρέπει να κινηθεί μια διαδικασία επί παραβάση βάση της συνθήκης λόγω του θέματος αυτού. Κατά τη δική μου εντύπωση. Πρόκειται για μια διαδικασία επί παραβάση εν γέννη σε σχέση με την ε, με την μεταγραφή της οδηγίας α, για τα θέματα περιβάλλοντος. να ξέρω λοιπόν αν πρόκειται για το συγκεκριμένο θέμα ή αν είναι ένα γενικότερο θέμα και θα ήθελα να θέσω το ερώτημα μήπως η Κομισιόν θα θεωρούσε ότι θα ήταν χρήσιμο τουλάχιστον να ανασταλεί η διαδικασία σχεδιασμού όσο τρέχει αυτή η διαδικασία. Και το τρίτο θέμα, έχουμε στην τσεχική δημοκρατία το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι τον Οκτώβριο, το προηγούμενο Οκτώβριο τροποποιήθηκαν οι κανόνες του παιχνιδιού μέχρι τον Οκτώβριο ήταν αρμόδια η κεντρική κυβέρνηση για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά από τον Οκτώβριο έχει μεταφερθεί αυτή η εξουσία στις περιφερειακές αρχές. Εγώ διαβάζοντας απλώς την ε, αναφορά, δεν ξέρω τα πραγματικά στοιχεία, αλλά ουσιαστικά έχει δώσει την έγκριση η κεντρική αρχή για αυτό το σχέδιο, ενώ βλέπω ότι οι περιφερειακές αρχές είναι εναντίον αυτού του σχεδίου. Μπορεί να υπάρχει λοιπόν μια τέτοια αντιπαράθεση και μήπως είναι αυτός ένας περαιτέρω λόγος για να υπάρξει επανεξέταση του θέματος αυτού και να ανασταλεί η διαδικασία. Τελευταίο ερώτημα προς την Κομισιόν. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξασφαλίσει ότι οι περιοχές προστασίας βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και από την γερμανική και από την τσεχική πλευρά να παραμείνουν προστατευμένοι ώστε αυτό το σχέδιο δεν θα βλάψει αυτές τις περιοχές. Αυτά λοιπόν και θα ήθελα να ενδεχομένως να επεκταθώ και στη συνέχεια. Τώρα, όταν εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζουμε να έχουμε περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας και είναι πολύ σημαντική αυτοί οι χώροι, Natura 2000 κτλ. θεωρώ ότι δεν μπορούν να συνδυάζονται αυτοί οι χώροι προστασίας με αιωλικά πάρκα ή υπάρχει κάποια διαφορετική αντιμετώπιση από την πλευρά της Κομισιόν. Αυτή είναι λοιπόν είναι η βασική αντιπαράθεση η οποία διαφαίνεται και από την αναφορά. Δεν ξέρω κατά πόσο η Επιτροπή θέλει να απαντήσει στις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε σχέση με τη διαδικασία επί παραβάση, όπως σας είπα, η Επιτροπή δεν μπορεί να εκκινήσει μια τέτοια διαδικασία ε, σε αυτό το στάδιο, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Εάν η Επιτροπή επιβεβαιώσει τις αντιρρήσεις των αναφερόντων, τότε θα μπορέσει να ζητήσει από τις τσεχικές αρχές να ε, γνωμοδοτήσουν ως προς τη μέχρι τώρα ακολουθούμενη διαδικασία. Επειδή η διαδικασία ε, πιστοποίησης ή αδειοδότησης χρειάζεται τουλάχιστον ένα χρόνο, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εκκινήσει μια διαδικασία επί παραβάση κατά των τσεχικών αρχών. Σε σχέση με την εφαρμογή της σχετικής οδηγίας, η Επιτροπή παρακολουθεί την υπόθεση εδώ και αρκετά χρόνια και δεν διαπίστωσε καμία παρέκκληση της διαδικασίας. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια διαδικασία που έχει διασυνοριακό χαρακτήρα ξεκίνησε από τις ε, περιφερειακές αρχές όταν ορίστηκαν και όταν ορίστηκαν αυτές οι διαστάσεις τότε η ανώτατη αρχή της ε, τσεχικής ε, δημοκρατίας δηλαδή το Υπουργείο Περιβάλλοντος ήρθε σε επαφή με τους ομολόγους από τη Γερμανία. Από αυτή την άποψη η Επιτροπή δεν διαπιστώνει διαδικασία παράβασης γενικότερα ως προς την εφαρμογή της οδηγίας σε σχέση με το, θέμα της ε, εμβέλειας θεωρούμε ότι υπάρχουν αρκετοί όροι που πρέπει να πληρούνται και γι' αυτό η διαδικασία θα επανεκκινήσει όταν πληρούνται αυτοί οι περιβαλλοντικοί όροι. Υπ' αυτή την έννοια, ελλείψη στοιχείων δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε παράβαση. Μιλάμε για ειδικά προστατευμένες περιοχές και θεωρούμε ότι το δίκτυο της τσεχικής δημοκρατίας επαρκεί για τους στόχους διατήρησης που ορίζονται από την οδηγία. Σας ευχαριστώ. Έχετε το λόγο. Επειδή η διαδικασία είναι εν εξελίξη, εγώ προτείνω να κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή. Βλέπουμε το πρόβλημα αυτό το οποίο συμβαίνει όταν έχουμε ήδη την έγκριση για το σχέδιο να προχωρήσει και από την άλλη πλευρά έχουμε παράπονα τα οποία διατυπώνονται. Μετά, αν αφήσουμε τα πράγματα να προχωρήσουμε, τότε θα έχουν δημιουργηθεί τα αεολικά πάρκα και το παράπονο δεν θα έχει κανένα, πρόβλημα, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Αλλά είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει σαν Επιτροπή Αναφορών τι κάνουμε όταν υπάρχουν σχέδια διαμεθοριακού χαρακτήρα για να συμμετέχουν και τα δύο εμπλεκόμενα κράτη. Είναι μια διαδικασία λοιπόν η οποία δεν επαρκεί σε αυτή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να σκεφτούμε στο μέλλον επομένως με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους θέματα. Γιατί δεν νομίζω ότι μπορούμε αλλιώς να βρούμε ικανοποιητικέ λύσεις. Παρακαλώ λοιπόν την Κομισιόν να παρακολουθήσει από πολύ κοντά το σχέδιο αυτό. Γιατί όταν έχει δοθεί ήδη η άδεια για την δημιουργία του αιωλικού πάρκου, το παράπονο το οποίο διατυπώνει και οι διαμαρτυρίες δεν έχουν πια κανένα αντικείμενο. Και κύριε Γιάρ, ε, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι η αναφορά αυτή προέρχεται από το δήμαρχο της περιοχής και επομένως ουσιαστικά είναι εκπρόσωπος της, ε, της περιοχής. Αλλά δεν προβλέπεται από την νομοθεσία η Κομισιόν να εξετάσει αυτές τις διαδικασίες ή να παίξει κάποιο διαμεσολαβητικό ρόλο. Και φυσικά η Κομισιόν η Επιτροπή μας θέλει να είναι κοντά στους πολίτες και να τους βοηθάει. Θα αφήσουμε λοιπόν ανοιχτή αυτή την αναφορά όπως προτείνει ο κ. Γιάρ και θα ζητήσουμε από τους ε, αναφερόμενους να μας πληροφορήσουν για τα συγκεκριμένα αιτήματά τους σε σχέση με αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, στην αρχή της συνεδρίασης είχαμε πάρει την απόφαση οι επόμενες ε, αναφορές, οι οκτώ και οι εννέα να εξεταστούν και κλεισμένων των θυρών. Θα δώσω λοιπόν ε, δύο λεπτά για να αποχωρήσουν όλοι εκτός από τους ε, έχοντες δικαίωμα να παραμείνουν. Μπορούν να παραμείνουν μονάχα αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό, οι βουλευτές, οι βοηθοί τους και από την Κομισιόν το άτομο το οποίο θα δώσει απάντηση σε σχέση με τις αναφορές υπαριθμών 8 και 9. Όλοι οι άλλοι παρακαλώ να φύγετε και πρωτού φύγουν θέλω να δώσω το λόγο στους δύο οι οποίοι θέλουν να λάβουν το λόγο. Ευχαριστώ. Όπως σας είπα, είχα αντιταχθεί στο να διενεργηθεί η συνεδρίαση και κλεισμένων των, ε, των θυρών. Οι αναφέροντες είναι παρόντες και θα ήθελα να λάβουν το λόγο και έχουμε και τρεις Σλοβάκους πολίτες ε, οι οποίοι δεν διαθέτουν, δεν τους ε, δόθηκε η ηθαγένεια. Θα ήθελα λοιπόν να μπορέσουν να παραμείνουν. Ε, θα ήθελα λοιπόν να απαντήσω το εξής το συναδελφός προς το πρώτο θέμα το σύστημα και των ε, θυρών θα ισχύει όπως ισχύει και στην περίπτωση που είναι δημόσια η ακρόαση. Θα δώσουμε το λόγο στους αναφέροντες στην Επιτροπή και μετά θα γίνει η ανοιχτή συζήτηση και οι αναφέροντες θα έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν. Εάν τα τρία αυτά πρόσωπα είναι αναφέροντες, τότε θα τους δώσω το λόγο θα μπορέσουν να λάβουν το λόγο. Μην ανησύχετε. Μου, ζήτησε το λόγο Είμαι, είμαι ο κύριος Τέκες. Κύριε Τέκες, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε. Την προηγούμενη Παρασκευή στείλαμε μια αίτηση προς την Προεδρία της Επιτροπής Αναφορών ε, με το όνομα της Άγνες Χόκες ε, Τύρκης Ορταμπόγκου ζητώντας να υπάρξει ανοιχτή συζήτηση. Ποια είναι η δικαιολογία της ε, συνεδρίασης και κλεισμένων των θύρων. Εγώ δεν καταλαβαίνω εδώ, δεν υπάρχει κάποιος κανονισμός που διέπει αυτό το θέμα. με κάθε σεβασμό θα σας απαντήσω για το θέμα αυτό. Το θέμα αυτό συζητήθηκε καταρχήν από την συνέλευση των συντονιστών όπου ελήφθη μια απόφαση. Και δεν υπήρξε κανείς ο οποίος ήταν εναντίον στην συνεδρία των συντονιστών. Όταν ξεκινήσαμε τη συνεδρίασή μας υπήρξε συζήτηση, πολλοί συνάδελφοι έλαβαν το λόγο, είπαν δεν συμφωνούμε με το να γίνει συζήτηση και κλεισμένο των θυρών. Γι' αυτό. Αν θέλετε, ζήτησαν πολλοί να γίνει μια ψηφοφορία για το να γίνει με ανοιχτό τρόπο η συζήτηση. Έγινε η ψηφοφορία, εσείς δεν ήσασταν παρόν, έγινε η ψηφοφορία και η ψηφοφορία κατέδειξε ότι η πλειοψηφία θέλαν να διατηρήσουν την κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίαση. Αν ήταν και ανοιχτών των θυρών συνεδρίαση, αν είχε επικρατήσει αυτή η άποψη, εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν προέδρευα τότε, ήταν η κυρία Ματσόνη η οποία προέδρευε, αλλά ήμουν δίπλα τη και μπορώ να σα διαβεβαιώσω και μπορώ να σα το διαβεβαιώσουν και οι συνάδελφοι ότι η ψηφοφορία κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό και υποστηρίζει επομένω την θέση των συντονιστών. Η, η κυρία εκεί πίσω, δεν μπορώ να δω το όνομά σας, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εάν οι συντονιστές αποφασίσουν ότι από τον επόμενο μήνα θα γίνονται αυτές οι συναντήσεις και κλεισμένων, εντάξει. Αλλιώς αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους χιλιάδες κανόνες με τον κανονισμό. Είναι αυθαίρετο. Τελείως αυθαίρετη η απόφαση. Ε, λέμε τόσα και τόσα για την διαφάνεια στην λήψη των αποφάσεων. Πώς είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι έχουμε και αυτές αξίες και αυτές οι αξίες να αγνοούνται. Έτσι, πρόκειται να αυτοχαρακτηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ως αφαίρετη πρόεδρος. Θα συμφωνούσα μαζί σας. Αλλά κρίμα γιατί εγώ δεν είμαι συντονιστή της ομάδας μας. Σε παρακαλώ Χριστίνα σηκώνει μια, μια κάρτα μεγάλη διαφάνεια η ομιλήτρια. Παρακαλώ, άστο, άστο. Οπότε, καλύτερα να έρθει σε επαφή με τον συντονιστή σου για το θέμα. Τώρα δεν μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα αυτό ήδη έχει συζητηθεί και ήδη έχει κρυθεί. Θα δώσω για δύο μόνο λεπτά στου συναδέλφου που έχουν ζητήσει το λόγο. Για δύο λεπτά μόνο. Θα ήθελα να, πούμε, να δούμε κάτι συγκεκριμένα ότι τον Μάρτιο που συνεντήθησαν οι συντονιστές επρόκειτο για μια αναφορά, μια άλλη αναφορά επί της οποίας αποφάσισαν οι συντονιστές ότι θα πρέπει να γίνει συνεδρίαση και κλεισμένο τρόπο Έχουμε άλλη αναφορά, αφορά τη διπλή ηθαγένεια, ε, υπευλήθη δύο μήνες αργότερα στην Επιτροπή μας. Οπότε, και ε, θεωρώ ότι η απόφαση των συντονιστών αφορούσε την πρώτη περίπτωση. Αυτή την απόφαση μπενά. Επ' αυτού έκριναν ότι θα πρέπει να γίνει συνάντηση και κλεισμένα και όχι επί της Δευτέρας περιπτώσεως. Γιατί τότε που ήρθε απόφαση των συντονιστών δεν είχε καν υποβληθεί η αναφορά και διπλή θα γίνει. Η επομένη ομιλήτρια. Πρόεδρε, αυτοί που συζήτησαν και απεφάσισαν για τη συνεδρίση και κλεισμένα δεν καταλαβαίνουν ότι για άλλη μια φορά εδώ έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν εδώ και μήνες επικρίθηκε σφόδρα η Ουγγαρία, είχαμε τότε την έκθεση Ταβάρες. Η έκθεση αυτή συζητήθηκε σε κάποια άλλη κοινοβουλική επιτροπή και επικρίθηκε η χώρα διότι ενεργούσε κατά τρόπο αντισυνταγματικό αλλά και προκειμένου. Δεν διαφέρει πολύ η περίπτωση. Και προκειμένου έχουμε συνταγματικό θέμα. Ε, τα περιεχόμενα σαν αναφορά επιδρούν στην κατάσταση των ποινών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν καταλαβαίνω ποια είναι η διαφορά. Γιατί θέλουμε ε, τώρα την συνεδρίαση κυκλισμένη. Γιατί δηλαδή να, να δίνεται δημοσιότητα στην υπόθεση Ταβάρες ενώ εν προκειμένου να εξαιρούμε, να αποκλείουμε τη συνεδρίαση τον κόσμο, να μπορεί να μπει στην αίθουσα και να γίνεται κυκλισμένο ο πρόεδρος. Εάν τώρα ανοίξουμε συζήτηση, θα στήσουμε τον κύριο Πέζη που περιμένει έξω. Ποιος μου περιμένει. Ε, στις 5.30 θα πρέπει να αρχίσει η νέα σύνδεση των συντονιστών. Παρακαλώ, να όσο πιο σύντομη μπορείτε, κύριε. Με την ευκαιρία που μου δίνετε, πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλοί θέλουν να γίνει ανοιχτή η συνδρίαση, αλλά ψηφίσαμε στην αρχή της, ε, της ημέρας. 9-4 εκρήθη θα έχουμε συνεδρίες και κλεισμένο. Σταματήστε να ε, χρησιμοποιείτε αυτή την υπόθεση για μικροπολιτικά συμφέροντα. Αλήθεια αυτό λέει ο Πρόεδρος. Όντως, δυστυχώς συμφωνώ. Στην αρχή της ημέρας έγινε ψηφοφορία με το δεδομένο αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι το οποίο αντιβαίνει στην ε, ε, απόφαση που έλαβε η Επιτροπή. Αυτό είναι το, το, το κυρίαρχο η ψηφοφορία και τα αποτελέσματά τη. Ε, αυτοί που ήθελαν κάτι άλλο θα μπορούσαν να είναι εδώ, θα μπορούσαν να έχουν ψηφίσει και να γύρει πλάστικα προς την άλλη μεριά. Θα κάνουμε ένα δίλεπτο διάλειμμα και συνεχίζουμε με τα σημεία 8 και 9.